Okay, So, uh, Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Φαίνεται ότι κάποιοι από εσά είναι τόσο εξαντλημένοι που δεν έχουν καν έρθει. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ ενδιαφέροντα σημεία στη μέση διάταξη σήμερα και με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τον καθηγητή Τσέλκε στην Επιτροπή μας. Και έχουμε και τον Τόμας ε, Σπένσερ, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ήταν ο Έλμαρ Μπρόκ της δεκαετίας του 80 ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Έχουμε προσκαλέσει τον καθηγητή Τσέλκε για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τις δια... δυνατότητες χρησιμοποίησης του πρωτοκόλου του Μοντρεάλ για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί μιλάμε πάντα στην Επιτροπή μας για το πρωτόκολλο του Κιώτο και το δεύτερο πρωτόκολλο του Κιώτο και είχαμε την Υπουργό Εξωτερικών του Μεξικού, την ε, κυρία Εσπινόζα που είναι η πρόεδρος του ΚΟΜ 16 και τις υποβάλλαν προτάσεις. Ποια είναι η άποψή σας για το κιότο 2 και έχουμε ξεχάσει ότι υπήρχε και πριν από το πρωτόκολλο του ΚΙοτο, το πρωτόκολλο του Μορεάλ και είναι κάτι το οποίο το παραγνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο και ότι μας δίνει κάποιες δυνατότητε για να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας κύριε Τσέλκε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να μας δώσετε ένα μήνυμα το οποίο θα μεταλαμβαδεύσουμε και στους άλλους συναδέλφους της ε, Επιτροπής μας. Ο καθηγητής Τσέλκε είναι ο επικεφαλής και ο ιδρυτής του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση στη Washington και στην Γενέβη και γραμματέας για την Διεθνή Γραμματεία για την συμμόρφωση και ε, επιβολή στα θέματα του περιβάλλοντος. Και έχει και σε διάφορα πανεπιστήμια διάφορες θέσεις. Δεν πρόκειται να σας τα αναφέρω όλα αυτά, θα πάρουν πολύ χρόνο. Έχετε το βιογραφικό του στο φακελό σας. Χαίρομαστε λοιπόν που είσαστε πάλι μεταξύ μας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να κάνετε αυτή την παρουσίαση και σίγουρο είμαι ότι τα μέλη μας θα έχουν ε, ερωτήσεις για να χρησιμοποιήσουμε τη μία ώρα που έχουμε για να εξετάσουμε τις δυνητικές ευκαιρίες που μας παρέχει το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι ευχαρίστηση που είμαι ξανά εδώ πέρα. Πάρα πολλά πράγματα συνέβησαν από όταν το ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα τον Ιούλιο. Εγώ χαίρομαι να έρχομαι στις Βρυξέλλες πάρα πολύ γιατί ως κάποιος ο οποίος περνάει το μισό του χρόνου στην Ουάσιγκτον χρειάζεται να έρχομαι εδώ για να έχω κάποια αίσθηση ευαισθησίας και αισιοδοξία για το κλίμα και μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα ακόμη περισσότερα μπορώ να σας πω. Πάντα λοιπόν χαίρομαι που έρχομαι εδώ. Το θέμα που θέλω να αναπτύξω σήμερα ξεκινάει με την υπενθύμηση πως η κλιματική αλλαγή είναι ακόμη δυσκολότερη ως προς την επίλυσή της μετά τα όσα έγιναν ε, στην Ιαπωνία, την τραγωδία στην Ιαπωνία. Ε, αξιολογούμε ξανά το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας και θα καθυστερήσουμε και θα ακυρωθεί σε πολλά μέρη. Αυτό το οποίο κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, η Κίνα για να αξιολογήσει δηλαδή τον κίνδυνο ασφαλείας θα αλλάξει το πως κοιτάμε τα πράγματα. Παρενθετικά όταν ήμουν νέος δικηγόρος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, είχα ασχοληθεί με την ποινική πτυχή του ατυχήματος στο Three Mile Island. Τα νέα από την Ιαπωνία φοβάμαι πως είναι πολύ χειρότερα μάλλον θα δούμε πως η τραγωδία αυτή είναι πολύ χειρότερη. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό, αλλά δεν ε, θα μου κάνει εντύπωση. Ταυτόχρονα είναι σκληρότερο να λύσουμε την κλιματική αλλαγή και πιο επίγονη η ικανότητά μας να διακυβερνήσουμε ε, δοκιμάζεται στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Ε, δεν είναι τόσο στιφαρή όσο συχνά νομίζουμε και όσο χρειαζόμαστε να είναι. Τι θα γίνει όταν έχουμε ταυτόχρονες αντικτύπους του κλίματος από μουσώνες που θα αλλάζουν, περισσότερες πλημμύρες, ξηρασίες, θα λιώνουν οι παγετώνες, ε, πυρκαγιές τα δάση που θα είναι πιο μεγάλες από ό,τι έχουμε δει. Έχουν ξεκινήσει ήδη αυτά, βλέπουμε στο Πακιστάν φέτος, ε, στη Ρωσία, το είδαμε στην Αυστραλία. Οπότε είναι επίγουσα, επίγον το πράγμα. Αυτό το κόστος ήδη ανεβαίνει όσον αφορά τον αντίκτυπο και ανεβαίνει γιατί όσο ε, αποδεχόμαστε διοξείδιο του άνθρακα και τους λοιπούς παράγοντες ε, τόσο περισσότερο μετά θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε. Ε, το κόστος ανεβαίνει Εάν χάσουμε τον πάγο τα καλοκαίρια στην Αρκτική θα αρχίσουμε να απελευθερώνουμε μεθάνιο και διοξίδιο του άνθρακα από τις μόνιμα παγωμένες περιοχές ε, που δεν θα είναι πλέον μονίμως πάνω παγωμένες και θα έχουμε πλέον μια λυσίδα η οποία θα οδηγήσει σε περισσότερο λιώσιμο, περισσότερη θέρμανση και ένα φαύλο κύκλο. Το έγγραφο το οποίο μοιράσαμε δείχνει στο σχήμα 1 που το έκανα με τον Μάριο Μολίνα από το Μεξικό έναν από αυτούς που πήραν ε, το Νόμπελ, ε, το βραβείο Νόμπελ μαζί με τους ε, Κρούτσεν και Ρόμπεν για την προστασία του όζοντος από τους χλωριοθωράνθρακες. Βλέπετε στο σχήμα 1 πως η θέρμανση την οποία έχουμε ήδη είναι πάρα πολύ κοντά στο να οδηγήσει σε απότομες εξελίξεις. Ε, θα πάμε λοιπόν από την Αρκτική, Μαλάια λοιπά. Μπορούμε να σκοτώσουμε ε, το δάστο Αμαζονίου περιμένοντας ε, περιμένοντας να κοπεί. Οπότε πρέπει να δράσουμε τώρα και επιθετικά. Αλλιώς μπορεί να δούμε πως η ικανότητά μας να κυβερνήσουμε ε, μπροστά σε αυτούς τους αντικτύπους θα ε, παρασυρθεί και τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε την κλιματική αλλαγή. Την έχουμε τώρα και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οπότε θα ήθελα εγώ σήμερα να εστιάσω στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο την πλευρά του διοξιδίου του άνθρακα, για την μείωση αλλά και, στη, και σε άλλα αέρια. Πρέπει, έχουμε πει πως θα πρέπει να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς ε, από τις προβιομηχανικές εποχές και 1,5 βαθμό ε, ως πιο λογικό στόχο που 100 χώρες είπαν στην Κοπενχάγη πως θεωρούν πως είναι το μάξιμο που μπορούν να ανεχτούν. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για θέρμανση, μιλάμε για 1,5-2 βαθμούς μιλάμε για παγκόσμιο μέσο όρο, δηλαδή στην Αφρική μιλάμε για μια μισή φορές πάνω από το παγκόσμιο μέσο όρο. Στα Ιμαλάια δύο φορές, στην Αρκτική δυόμιση φορές το παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή η μέση όρη είναι παραπλανητική. Αν φτάσουμε στους δύο βαθμούς, άλλος ένας βαθμός δηλαδή για την Αφρική, και άλλοι δύο βαθμοί συν για τα, τα και την Αρκτική δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε αυτά. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, με τον ΟΗΕ, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά αντιλαμβανόμαστε πώς δεν είναι ο γρήγορος τρόπος για να επιτύχουμε περιορισμό. Και αν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία το πολύ είπαμε στην Κοπενχάγη, θα έχουμε 60% της μείωσης που χρειαζόμαστε μέχρι το 2020. Ε, μπορεί να πει κανείς ότι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι, ανάλογα πώς το βλέπει. Μισογεμάτο σημαίνει λίγο παραπάνω από μισογεμάτο. Εάν αυτή η συνθήκη έχει αυτό το ποσό, θα έλεγα πως είναι αρκετά καλό αποτέλεσμα για μία μόνο συνθήκη, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να δούμε και άλλους νόμους, θεσμικά όργανα, άλλους φορείς όπου μπορούμε να μειώσουμε πιο γρήγορα. Και όλοι αυτοί είναι, σχεδόν όλοι, εκτός του διοξιδίου του άνθρακα. Χρειαζόμαστε λοιπόν συμπληρωματικές δράσεις πλην του διοξιδίου του άνθρακα που θα αναλυθούν γρήγορα, να επιταχύνουν τα πράγματα. Είμαστε ήδη σε επικίνδυνες καταστάσεις και έχουμε αρχίσει και χτυπάμε στις μπαριέρες. Μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε κάποιες δράσεις. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι 50% ε, ε, έχει αυξηθεί 50% από το 1970, είναι το μεγαλύτερο στοιχείο και σε αυτό εστιάζουμε. Επίσης, ε, είναι επίμονο. Μένει δηλαδή στην ατμόσφαιρα ένα κομμάτι του για χιλιάδες χρόνια. Οι δε δυνάμεις μη διοξείδιου του άνθρακα έχουν μικρούς χρόνους παραμένουν στην ατμόσφαιρα από ώρες μέχρι μέρες, λίγες εβδομάδες, μέχρι κανένα δύο δεκαετίες. Δύο δεκαετίες είναι πολύ γρήγορο σε σχέση με τις χιλιετίες. Η αξιολόγηση που έγινε από το πρόγραμμα του περιβάλλοντος του ΟΗΕ, το Παγκόσμιο Μητρολογικό Οργανισμό, δείχνει πως μπορούμε να μιλάμε ε, να φτάσουμε στους δύο βαθμούς σε 60 χρόνια. Αν ε, εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα ε, ασχοληθούμε και με άλλα αέρια και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως εξασφάλιση. Μπορούμε να κόψουμε τις προσπάθειες να μειώσουμε το ρυθμό αύξησης στο μισό. Στη δε αρκτική κατά δύο τρίτα. Φοβερά πράγματα να μειωθεί ο ρυθμός θέρμανσης με το να προσθέσουμε τα αέρια που δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα. Η Αρκτική που έχει σημασία για την Ευρώπη και τον κόσμο, η Αρκτική είναι μια σπίδα προστασίας. Ο λευκός άσος αντανακλά τη ζέστη. Και αν αντικαταστήσουμε με μαύρο νερό, απορροφάται η ζέστη από του ωκεανούς και επιταχύνει τη θέρμανση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κόψουμε τη θέρμανση της Αρκτικής. Τώρα η ρήπη μη διοξιδίου του άνθρακα είναι υδροφθοράνθρακες που υπάρχουν στα ψυγή και διαλυτικά και έχουν άλλες χρήσεις. Αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης τη μούργα του άνθρακα που είναι ίσως ε, το σημαντικότερο, η καπνιά δηλαδή, το σημαντικότερο κομμάτι πλην του διοξιδίου του άνθρακα. Και βεβαίως υπάρχει και το μεθάνιο αέριο του θερμοκηπίου Αυτά είναι τα πλήν του διοξιδίου του άνθρακα και μιλάμε για γύρω στο 50% από το 1970. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους που μπορούν να μας κρατήσουν κάτω από τους δύο βαθμούς, να μειώσουν κατά δύο τρίτα το ρυθμό της θέρμανσης και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της υπάρχουσας νομοθεσίας και θεσμών και τεχνολογιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσουμε με τους ε, ή υδροφροναθρακής, με συγχωρείτε, είναι αυτοί που αναπτύσσονται ταχύτερα στη ΣΥΠΑ και αλλού. Οι 27 της Ένωσης έχουν αυξήσει τις εκπομπές τους ε, κατά 85% μεταξύ του 1990 και του 2008, ενώ τα υπόλοιπα 5 αεροθερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 14%. Είμαστε σε άσχημο δρόμο δηλαδή με τους υδροφροναθρακές. Εάν δεν αρχίσουμε να τους ρυθμίζουμε, θα συνεισφέρουν γύρω στο 50% του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Δηλαδή μιλάμε 13 χρόνια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σοβαρό πρόβλημα. Τα στοιχεία είναι στο έγγραφο του κυρίου Μολίνα. Εάν όμως τους ελέγξουμε... Now. Πάρα πολύ γρήγορα να μειώσουμε το ρυθμό θέρμανσης. Εάν η παραγωγή των στοιχείων αυτών έμπαινε στο ε, πρωτόκολλο του Μοντρεάλ μπορούμε να εξαφανίσουμε ένα από τα έξι αέρια του θερμοκηπίου. Όχι εμπόριο, μείωση, αγορά και τέτοια. Είναι είναι ένα συνθετικό, μια συνθετική ουσία την οποία εμείς κατασκευάζουμε και θα πούμε δεν την κατασκευάζουμε και θα πάμε σε άλλες εναλλακτικέ. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε εδώ πέρα. Τώρα το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Για όσους το ξέχασαν πόσο υπέροχο είναι, είναι η καλύτερη περιβαλλοντική συνθήκη που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Και οφείλω να συγχαρώ την Ευρώπη για το ότι επέδειξε ηγετικό ρόλο. Η συνθήκη αυτή κατήργησε σταδιακά 96 βλαβερές χημικές ουσίες κατά 98% μεταξύ του 1990 και 2010. 240 κλάδοι της βιομηχανίας κατά 96% κατά 98% σε 96 στοιχεία. Και έτσι θα ανακάμψει μέχρι το 2065 το στρώμα του όζοντος. Γιατί, ξέρετε, οι χλωροθωράνθρακες μένουν καιρό στην ατμόσφαιρα και βλάπτουν τη στρατόσφαιρα κτλ. Ταυτόχρονα, ενώ βρίσκεται σε καλό δρόμο το στρώμα του όζοντος, για εμάς ε, έχει, κάνει έχει βοηθήσει περισσότερο το κλίμα από οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για 135 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα. 11 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο. Είναι τρομερή συνεισφορά. Το συνολική τιμή που πληρώνει το κοινό μέσω του πολυμερούς ταμείου είναι 4 cents τον τόνο. Οπότε είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η συνθήκη. Δυστυχώ και ευθυνή η συνθήκη εννοούσα. Βεβαίω, πολλέ χώρε του κόσμου είπανε Α, καλή δουλειά έκανε αυτή η συνθήκη, τώρα δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό το θέμα στο μέλλον. Μπορούμε λοιπόν να πάει σιγά σιγά να πηγαίνει στο υπόγειο και να τελευταίσει το βίων. Ενώ δεν είναι το δικό μου αυτό το τηλέφωνο. Και να εξαντλήσει εκεί τη χρησιμότητά της. Αυτό όμως θα ήταν σοβαρό λάθος γιατί το πρωτόκολλο του Μονρεάλ μπορεί ακόμα να κάνει για το κλίμα όσα έχει ήδη κάνει. Αν κάνουμε αυτά τα πράγματα λοιπόν για τους υδροφθοράνθακες και τους χλωροφθοράνθακες τα έχουμε κάνει αυτά, μπορούμε να μειώσουμε με 5 ή 10 σέντ τον τόνο τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό μέτρο που μπορεί να γίνει μέσα από μια συμφωνία, μια διεθνή συμφωνία. Ναι, ναι, πρέπει να κάνουμε μερικά τελικά σχόλια γιατί περνάει η ώρα η προσπάθεια που έγινε για την αντιμετώπιση της τρύπα του όζοντος έχει επιλύσει ένα μείζον πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αν θυμάστε το παρελθόν ξεκίνησε αυτό με θελοντικές προσπάθειες αλλιώς το πρόβλημα αυτό θα ήταν εξίσου μεγάλη σοβαρότητα όπως το σημερινό πρόβλημα του διοξιδίου του άνθρακος. Επομένως σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του, του του περιβάλλοντος. Γιατί η τρύπα του όζοντος, όπως σας είπα προηγουμένως, οδηγούσε σε μια αύξηση της κατακρατούμενης ακτινοβολίας κατά 1,6 βάτο τετραγωνικό μέτρο. Έχουμε λοιπόν πολλές ε, μορφές ρήπων που είναι τοπικού χαρακτήρα η παρουσία τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες και εθνικούς και περιφερειακούς ε, νόμους για να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη δημόσια υγεία, σώζει 2,5 εκατομμύρια ζωές στον χρόνο που υποφέρουν από την καπνιά του μαύρου άνθρακα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρύπα του όζοντος. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο μέρος του μηνύματός μας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη με όλα αυτά. Εντάξει, είμαι διαθέσιμος να το συζητήσω μαζί σας. Αλλά οι χώρες BRICS, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Κορέα, όλες αυτές οι χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν και πρέπει να το κάνουν σύντομα θα κλείσω εδώ προς το παρόν κύριε Πρόεδρε και είμαι έτοιμος να απαντήσω ερωτήσεις. Yeah, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και για τα τόσο εντυπωσιακά στοιχεία που μας αναφέρατε. Είναι πράγματι εντυπωσιακό και εκπληκτικό το ότι το πρωτόκολλο του Μορεάλ δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους μας. Τι κάνει όμως το Διεθνές Πάνελ για την κλιματική αλλαγή, το IPCC του ΟΗΕ. Γιατί θα πρέπει να καλύψει τη συνολική εικόνα για το περιβάλλον και όχι μοναχά το θέμα του διοξίδιου του άνθρακος. Εγώ δεν ξέρω όμως ακριβώς τι έχει κάνει το Διεθνές Πάνελ για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ένα άλλο ερώτημα Αναφερθήκατε στους υδροφθοράνθρακες. Εξετάσαμε αυτό το θέμα με το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Ο στόχος ήταν να καταστραφούν αυτοί οι υδροφθοράνθρακες με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες παρήγαγαν λίγο περισσότερους τέτοιους ε, υδροφθοράνθρακες για να πάρουν πιο πολλά λεφτά από το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Και εσείς μας είπατε ότι από το 1990 έχει αυξηθεί σημαντικά η παρουσία αυτών των υδροφθοροανθράκων. Είναι όμως μέσα στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ή όχι, θα ήθελα να απαντήσετε. Και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα συνάδελφοι, ίσως μπορούμε να συνενώσουμε δύο-τρία ερωτήματα για να τα απαντήσετε από κοινού και ομού ο Θεόδωρος Σκυλακάκης. thank you for coming here and... Ευχαριστώ που ήρθατε και που μας ανοίξατε τα μάτια. Μερικές φορές δεν βλέπουμε το προφανές στην πολιτική. Και νομίζω πως ε, αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Δύο ερωτήσεις έχω. Εγώ παρακολουθώ το ζήτημα των ε, υδροφθορανθράκων ε, και προσπαθώ να κινητοποιήσω τον κόσμο να βγάλει το HFC-23 από τον καθαρό, μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης γιατί είναι παρανοϊκό να πληρώνουμε με 12 και 14 δολάρια κάτι το οποίο γίνεται με 17 cents. Και το καταφέραμε αυτό με, την, με τη βοήθεια συναδέλφων το επιτύχαμε αρκετά γρήγορα. Έφυγαν λοιπόν, έφυγε το HFC 23 που είναι αρκετά σημαντικό αέριο από μόνο του. Αλλά είναι τώρα εκτός γενικώ, δεν καλύπτεται από τίποτα. Κάτι το οποίο δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή γιατί έτσι μπορεί να επικεντρώσουμε την προσοχή κάπου, γιατί μέχρι τώρα οι παραγωγοί είχαν δυνατότητα να κερδίσουν τόσο τεράστια ποσά που μπλοκάριζαν το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Οπότε έπρεπε να το βγάλουμε εκτός για να ανοίξει ο δρόμος για το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ και τους ε, υδροθονάνθρακες ε, συνολικά. Ε, ε, βεβαίως έκανα την ίδια ερώτηση νησιών ε, τον Οκτώβριο και βεβαίω υποστηρίζω ε, να λύσουμε το ζήτημα του κλίματος μέσω των ε, υδροφθοναφρακών. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διμερέ και να αγοράσουμε φτηνά π.χ. το HFC 23 το οποίο δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο του Μονρεάλ γιατί δεν ευλάπτει το όζον και να δείξουμε στον κόσμο πως είναι σοβαρό το θέμα και κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση και την έχω απευθύνει και στην Κομισιόν τον Σεπτέμβριο. Αλλά έπρεπε να το αφαιρέσουμε αυτό πριν γίνει οτιδήποτε. Τώρα νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο από την προσπάθεια να πάμε από το διοξείδιο του άνθρακα το 20 στο 30 στην Ευρώπη. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η Ευρώπη μπορεί να τα αγοράσει αυτό. 20% εάν ε, προχωρήσουμε ε, προς τα εκεί. θα έχει έτσι πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας πως η κλιματική πολιτική έχει μπει στην πολιτική τη γενικότερη. Και ο καθένας έχει αυτό που του αρέσει. Ε, ηλιακά πάνελ, ε, δάση, αρκτική, διάφορα. Ο καθένας έχει το αγαπημένο του. Και με τον ασχολείο το καθένας με το αγαπημένο του ξεχνάμε το, το βράκο αν θέλετε, με το αγαπημένο του ζωάκι. Και ο μπαμπούλα είναι εδώ. Και θα μας φάει. Και πρέπει να επικεντρωθούμε με αποτελεσματικούς τρόπους ε, αντιμετώπισης του. Αν ήξερε ο κόσμος ότι ξοδεύουμε 15 δολάρια ενώ μπορούμε να ξοδεύσουμε 5 cents δεν ε, δεν θα ξεμπλέκαμε εύκολα. Και πριν το μάθουν καλύτερα, ε, ας πάμε να ξοδέψουμε τα 5 cents. Ευχαριστώ. Yeah, thank you, Ευχαριστούμε. Α, επομένως έχουμε μπροστά μας το τέρας αυτό. Και όχι μονάχα... Δεν έχουμε μονάχα παιχνιδάκια μόνα μας, έχουμε ενώπιό μας ένα δράκο. Η Κριστίνα Γκουτιέρες τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζέλκε για την παρουσία του. Υπάρχει κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Ίσως το βλέπω με θηλυκή λογική, αλλά μου φαίνεται ότι μερικές φορές το μικρό είναι σημαντικό. Και εδώ δεν συμφωνώ απόλυτα με τον ε, κύριο Σκυλακάκη. Εγώ πιστεύω ότι για την κοινωνία το θέμα του πρωτοκόλλου του Μορεάλ, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το σύνολο αυτό λοιπόν το, της προβληματικής. Το θέμα της μείωσης των εκπομπών είναι ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο, τόσο αφηρημένο που ξεπερνάει την ανθρώπινη αντίληψη και φαίνεται αδύνατο να το αντιμετωπίσει ο κόσμος. Είναι, φαίνεται κάτι το οποίο μόνο τα κράτη, τα κράτη του κόσμου, οι μεγάλες χώρες μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Έχουν περάσει λοιπόν πολλά χρόνια. Δεν λειτουργεί η μετάφραση. Δεν λειτουργούν τα μηχανήματα, κύριε καθηγητά. Μετάφραση. Α, εντάξει, καταλάβατε τώρα, εντάξει. Ξαναρχίζω. Μου δίνεται, μου δίνεται λοιπόν η εντύπωση, επειδή είμαι και καθηγήτρια στο κάτω-κάτω, ότι στην κοινωνία μας η έννοια της κλιματικής αλλαγής σαν σύνολο, Μοντρεάλ, Κοπενχάγη, Κανκούν, Όλα αυτά δημιουργούν τόσο μεγάλο και τόσο αφηρημένο πρόβλημα για τον κόσμο που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και αιώνες θα έλεγα, εμείς εναποθέτουμε στα κράτη αυτό το οποίο έπρεπε να είναι ατομική ευθύνη και την ελπίδα να λύσουν τα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι η έλλειψη κατανόησης και η αδυναμία να κάνουμε μια ριζική αλλαγή στα, στις συνήθειές μας είναι κάτι πολύ δύσκολο για μια κοινωνία που θεωρεί ότι αυτό το εγχείρημα είναι κάτι το τεράστιο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να παίξουμε και ένα παιδαγωγικό ρόλο. Και πιστεύω ότι τα μικρά μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα λίγα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς από το σπίτι του, από την αυλή του, από το δήμο του. Μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το γενικό φαινόμενο. Μόνο έτσι μπορεί να υπε... υπευθυνοποιηθεί η κοινωνία. Ξέρουμε ότι ένα παιδί δεν μαθαίνει κάτι άμα δεν το κάνει το ίδιο. Δεν μπορούμε να μάθουμε ένα παιδί να μαγειρεύει άμα δεν το κάνει μόνο του. Όλα τα πράγματα πρέπει να περάσουν από την πρακτική. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν ώστε να υπάρχει αυτή η γενική πρακτική και κάνοντας κάτι το ερωτεύεται κανείς στο τέλος. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την πολιτική κίνηση οι, επιστημόν, οι επιστημόνες, επιστήμονες πρέπει να βοηθήσουν την κοινωνία να κόψει το πρόβλημα αυτό σε μικρά κομμάτια που να είναι επιλύσιμα. Η πρόταση τώρα της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας να αρχίσουμε να εργασόμαστε σε συγκεκριμένους τομείς της κλιματικής αλλαγής. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ σημαντική, γιατί πέραν των γενικών στόχων που έχουμε διατυπώσει στην Κοπενχάγη. Αν κάθε τομέας έχει μια χωριστή υπευθυνοποίηση, δεν θα έχουμε προβλήματα ανταγωνισμού. Αντί να δώσουμε μια πανάκια, μια λύση για όλα τα επίπεδα, να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες εναλλακτικέ λύσεις που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες λύσεις ανά τομής. Και έτσι να συνενώσουμε τις προτάσεις για τους μεγάλους στόχους σε οικουμενικό επίπεδο που υπογράφουν τα μεγάλα κράτη στον κόσμο μας με προτάσεις πιο συγκεκριμένες για διάφορους τομείς και για διάφορες ομάδες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια δημοτική πολιτική ανάπτυξης, μια δημοτική πολιτική για τον άνθρακα, μια πολιτική δημοτική ακόμα και για τη Γεωργία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτά τα οποία είπε ο κύριος καθηγητής ήταν ενδιαφέροντα. Αναρωτιέμαι μόνο γιατί η διεθνής κοινότητα δεν πάει στην κατεύθυνση την οποία μας είπατε. Γιατί από όσο ξέρω νομίζω το να ζούμε χωρίς ε, αυτά τα αέρια είναι πολύ απλό και δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά. Ενώ αυτό το οποίο έχουμε διαλέξει τώρα να ακολουθήσουμε σημαίνει τεράστιες ε, μεταβολές. Δηλαδή αν είναι να ασχοληθούμε ε, μόνο με την ε, κλιματική αλλαγή, εντάξει είναι φιλόδοξος ο στόχος για το διοξίδιο του άνθρακα, και μέχρι το 2050 θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, ούτως ή άλλως, εντάξει, για λόγους σπόρων, αποτελεσματικότητας κτλ. Αλλά όσον αφορά μόνο την κλιματική αλλαγή, αναρωτιέμαι γιατί η ενταξει για λογους σπορων αποτελεσματικοτητας κτλ αλλα οσον αφορα μονο την κλιματικη αλλαγη αναρωτιεμαι γιατι η κοινοτητα και η επιστημονική κοινότητα δεν ασχολήθηκε με τη δεύτερη πτυχή που μας αναφέρατε μόλις τώρα, γιατί αν κατάλαβα καλά είναι ε, πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτός, χωρίς μεγάλα πολιτικά προβλήματα. Τρίτον, με το πρωτόκολλο του Μονρεάλ, έχουμε ε, ήδη κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα με μια παγκόσμια συνθήκη. Και είπατε και εσείς πως είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί δεν καταφέρνουμε λοιπόν να συμπληρώσουμε αυτή τη συνθήκη για να καλύψουμε τις πτυχές του κλίματος εφόσον έχουμε ήδη σε ένα μέρος μία συμφωνία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν γιατί ούτε από πολιτική ούτε από επιστημονική σκοπιά δεν ε, κινηθήκαμε προς τα εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της παρέμβασής του. Είπατε, το μικρόφωνο δεν λειτουργεί το μιλτή. Λοιπόν, Κύριε καθηγητά, είπατε στην αρχή της εισήγησής σας ότι λόγω των γεγονότων στην Ιαπωνία θα υπάρξει μείωση στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Είπατε επίσης, και αυτό είναι μια γενική προσπάθεια, ότι χρειάζεται να περιοριστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει περιορισμός της παραδοσιακής παραγωγής, των παραδοσιακών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει αύξηση στη ζήτηση ενέργειας στην ε, Κίνα και αλλού. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. χρησιμοποιούμε όσο, όλο και λιγότερο πετρέλαιο, όλο και λιγότερη πυρηνική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη ενέργεια. Πώ μπορούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε την έλλειψη αυτή και με τι κόστο. πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε συχνά, έχετε αναλύσει τον αντίκτυπο της αύξησης του πληθυσμού στις κλιματικές αλλαγές. Γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η όγκη όλων των αγαθών που χρειαζόμαστε και καταναλώνουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα εδώ να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά έχετε σκεφτεί τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή αύξηση του πληθυσμού και κλιματικών αλλαγών. Any other Άλλες παρεμβάσεις, ο Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη συνέχεια των σχολείων του κυρίου Σίμπερ, όσον αφορά την ανταπόκριση από την Κομισιόν στο έγγραφο και στις προτάσεις που περιέχει αυτό, είναι μια λίστα με πράγματα που θα πρέπει να γίνουν ώστε να συμβούν στη συνέχεια όλα αυτά. a few questions. Okay. Έχετε λοιπόν μερικέ ερωτήσει. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες απαντήσει, σα δούμε. Στην αρχή, για τον πρώτο κύριο που μίλησε, σίγουρα συμφωνώ με την παρουσίαση των ε, θεμάτων ε, για το HFC 23. Έχουμε, είναι όντω αλήθεια ότι πληρώνουμε υπερβολικά μεγάλα ποσά για αυτά τα προϊόντα και έτσι έχουμε δημιουργήσει κίνητρα για να καθυστερήσουμε την περαιτέρω χρήση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τους, ε, για τους υπόλοιπους ε, υδροφθοράνθρακες και τους χλωροφθοράνθρακες και για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούμε το HFC 23. Αν περιορίσουμε περισσότερο το HFC και το βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο πρωτόκολλο που να λειτουργεί ταχύτερα, νομίζω πως θα προχωρήσουν καλύτερα τα πράγματα. Η ιδέα σας για τη δημιουργία διμερών ε, ταμείων θα ήταν εξαιρετική ιδέα και είναι πολύ φθηνές πιστώσεις. Η ερώτησή μου είναι πόσες από τις πιστώσεις από αυτές θα τις χρησιμοποιούσες για αναχέτηση και για, για αντικατάσταση και πώς από αυτά θα χρησιμοποιούσατε για να βγάλετε από την αγορά τελείως αυτά τα προϊόντα, ώστε να μην χρησιμοποιούνται εν καιρό. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ως πολιτική θα πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί η αναχέτηση μπορεί να σημάνει την καθυστέρηση της ιδέας, της χρήσης μάλλον των ε, προϊόντων αυτών. η Ισπανίδα βουλευτής μου ζήτησε να το σχολιάσω και είπε ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα έτσι όπω παρουσιάζεται που ο κόσμος παραλύει και τελικά δεν κάνει τίποτα. Είναι πολύ σημαντική ιδέα γιατί Εάν μοιράσουμε το κλιματικό πρόβλημα σε, τοπικές, σε τοπικά κομμάτια, ίσως να βρούμε πιο ευφυείς λύσεις. Και ακριβώς αυτό έκανε και το πρωτόκαλο του, Μόντρεαλ. Αν απεικοδομήσουμε το, τη συνθήκη, φτάνουμε σε 23 χρόνια πριν, που, όπου είπαμε βγάζουμε τα αέρια του θερμοκηπίου και θα φτιάξουμε μια ειδική συνθήκη, κομμένη και ραμμένη, ώστε να ξεφορτωθούμε αυτά τα χημικά. Και έγινε πολύ καλή δουλειά. Αρχίσαμε τα, με μικρούς στόχους, μαθαίνουμε καθώς ε, προχωρούμε και έκτοτε έχουμε ε, καταργήσει 96 χημικές ουσίες. Συμφωνώ λοιπόν ότι περαιτέρω τομεακές προσεγγίσεις θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί τώρα η διεθνής κοινότητα ακόμα δεν ακολουθεί αυτή τη στρατηγική ώστε να συμπεριληφθεί η παραγωγή και η κατανάλωση των HFC στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Διάφορες χώρες το έχουν κάνει, κυρίως ε, οι νησιωτικές χώρες, Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, ο Μαυρίκιος, είπαν ε, ότι εμείς σήμερα ήδη υποφέρουμε από τις κλιματικές αλλαγές, χρειαζόμαστε πολύ γρήγορη ε, αναχέτηση ε, των, κλιματικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να επικυρωθεί μια συνθήκη και να εφαρμοστεί. Πρέπει σήμερα να δράσουμε. Και γι' αυτό και ε, οδήγησαν ε, το ΣΥΠΑ, Καναδά και Μεξικό να υποβάλουν πρόταση. Οι Ευρωπαίοι και οι Ιάπωνες υποστήριξαν αυτή τη λύση και πολλές άλλες χώρες, 91 χώρες μάλιστα, είπαν ναι, χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο για να ενεργήσουμε πιο γρήγορα και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Νομίζω λοιπόν πως είμαστε στο σωστό δρόμο ε, και επίσης υπήρξε μια μεγάλη σημαντική στιγμή όπου ο Υπουργός Ραμάστης Ινδία είπε ότι η... Η Ινδία μπορεί να ηγηθεί της ε, κατάργησης των HFC από τη στιγμή που υπάρχει υποκατάστατο είναι πολύ ευφυής πολιτικός. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τον βρούμε τη λύση για να τον βοηθήσουμε στο να υλοποιήσει αυτή την φιλόδοξη πολιτική δήλωση που έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Το σχόλιο μου για την πυρηνική ενέργεια. Εγώ νομίζω ότι ναι, μεν ο κόσμο μπορεί να συνεχίσει να λέει ότι θα φτιάξουμε τα πυρηνικά μα εργοστάσια όπω τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά τουλάχιστον θα υπάρξει κάποια, σταθερο... Ε, ε, κάποια καθυστέρηση και θα εξετάσουν περισσότερο την ασφάλεια. Και ίσω κάποιε χώρε να πούνε ότι μπορεί να μην είναι και τόσο τέλεια επένδυση. Κάποια δισεκατομμύρια κοστίζει η κατασκευή ενό πυρηνικού εργοστασίου και μπορεί να υπάρξουν προβλήματα που να κοστίσουν τρισεκατομμύρια δολαρίων. Αλλά ναι, χρειαζόμαστε ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια. Είναι ε, ένα θέμα, ένα πρόβλημα μάλλον, το οποίο απασχολεί όλους όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, γιατί έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αναπτύσσεται και χρειάζεται ενέργεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενέργεια και για την διατήρηση του περιβάλλοντος. Όταν χρησιμοποιούνται στερεά καύσιμα, θα πρέπει να σκεφτούμε την υποχρεωτική άμβληση των, ε, των επιπτώσεων. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αν επεκτενόταν η παραγωγή βιομάζας, αν ε, μετατρέπαμε τη βιομάζα μέσω πυρόλησης σε ε, σε κάποιες πιο συμπαγές, σε ένα είδος συμπαγούς άνθρακα. Σε λίγα χρόνια άλλα τρία δις ε, άνθρωποι προβλέπονται, προβλέπονται ότι θα ζουν πάνω στον τον ίδιο πλανήτη. Τεράστια πρόκληση. Καλύτερος τρόπος είναι να τους εκπαιδεύουμε. Είναι στρατηγική ανθρωπίνα δικαιωμάτων, στρατηγική για τα δύο φύλλα. Ε, είναι το να εκπαιδευτεί ο κόσμος, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο που δεν εκπαιδεύονται ε, τα παιδιά εκεί. Ο τελευταίο ομιλητή μου ζήτησε κατάλογο με τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ποιο θα ήταν το σωστότερο να κάνουμε τώρα. Καταρχήν, θα πρέπει η Ευρώπη να, δείξει, να παίξει ηγετικό ρόλο εδώ, να πρωτοπορήσει. Ε, στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη, μεγάλο κεφάλαιο γνώση όσον αφορά τι κλιματικές αλλαγέ. Στον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι τόσο προηγμένη η σχετική έρευνα. Ακόμα και σε συντηρητικέ εποχές είχαμε καλές εκθέσεις και στη ΣΥΠΑ με τον Ρόναλντ Ρέγκεν, με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Ε, υπάρχει θέμα χρηματοδότησης Φέτος οι χώρες δωρητές ε, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων θα πρέπει να ξαναγεμίσουν τα πολυμερή τους ταμεία, να βάζουν 500 δις δολάρια το χρόνο, 5 ε, ε, δις συγγνώμη το χρόνο και θα πρέπει μάλλον να βάλουμε άλλο ένα 50% αν θέλουμε δύο phase out να κάνουμε ταυτόχρονα. Ειδικά για τον άνθρακα η πρόταση αυτή είναι πολύ πολύ συμφέρουσα. Τα 5 cents το τόνο. Νομίζω λοιπόν πως κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι εφικτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυλακάκης θέλει είχε, βάλει, είχε θέσει μια ερώτηση και στην Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που μου έθεσε ο κύριος καθηγητής. Ποια είναι η γνώμη μου για τις πιστώσεις σε περιπτώσεις ε, διμερών συμφωνιών. Όχι, δεν θέλω πιστώσεις. Να αγοράσει κανείς ολόκληρο το εγχείρημα αυτό και να δώσει στον κόσμο 10-12% ε, απόδοση για τις επενδύσεις του. Να ξεχάσουμε τις πιστώσεις. Τι χρειάζεται να φτιάξεις. Έναν αποτεφρωτή ε, θα το βάλουμε εκεί, θα το φτιάξουμε, θα πληρώσουμε μέχρι το 2030 ή όσο καιρό, εν χρειαστεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει και θα, σου σας δώσουμε 10% απόδοση γι' αυτό. Και δίνουμε και τα χρήματα γι' αυτό όλα αυτά. Ας μας απαντήσει και ο Φίλιπ από την Κομισιόν, αν θέλει να παρέμβει για το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να παρέμβετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έσω έτοιμος βεβαίως, όπως λένε. Λοιπόν, Παρακολουθούμε τη συζήτηση αυτή πάρα πολύ στενά στο πρωτόκολλο του Μοντρεάλ. Όπως θα ξέρετε, επιδείξαμε ηγεσία στην τελευταία συνάντηση των μερών στην Μπαγκόγκ τον περασμένο Νοέμβριο που ε, φροντίσαμε από νωρίς να υποστηρίξουμε την πρόταση της Βορείου Αμερικής και της Μικρονησίας για να καταργηθούν σταδιακά εντός μιας 20 τα αέρια αυτά. Ήταν δύσκολες οι συζητήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και βεβαίως είχαμε δυσκολίες από τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα και στη τελική ανάλυση είχαμε λίγη πρόοδο, μικρή πρόοδο. Όμως, από την άλλη, όπως είπατε, είχαμε δηλώσεις που υπέγραψαν 91 μέρη, 27 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς καλά τα πήγαμε ναι, μεταξύ των 91 δηλαδή που υπέγραψαν από εδώ και μπρο. τι κάνουμε. Οπωσδήποτε στο Κανκούν ο Ινδό υπουργό είπε πω ε, γίνονταν εργαστήρια με τι ΗΠΑ ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό με τις ΗΠΑ έγινε στο Δελχή πριν από λίγες εβδομάδες και είμαστε σε επαφή με το επιτελείο του Υπουργού να δούμε πώς θα πρέπει να υπάρχει και μια ανάλογη συνάντηση και περιμένουμε. Στο μέλλον θα έχουμε μία ομάδα εργασίας για να προετοιμάσουμε την συνάντηση τον Αύγουστο που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο βεβαίως και αναμένουμε να δούμε τι θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αν υπάρχει νέα πρόταση για να μειωθούν ε, οι προφθοράνθρακες από τα συμβαλόμενα μέρη. Ευχαριστώ. Ο Κρίς, ναι, ένα σύντομο ερωτηματάκι. Είναι αλήθεια ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Όβεν, μήπως πράγματι αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Υπάρχει μια παράλληλη διαδικασία η οποία είναι εν εξελίξη, λέει ο κύριος Όβεν. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουμε μια σειρά από μελέτες οι οποίες είναι σε επεξεργασία. Και όταν τελειώσει αυτό το έργο θα δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε πώς θα κινηθεί η αγορά και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα αυτών των μελετών. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. αυτό είναι χωρίς το θέμα, λέει ο κύριος Ντέιβιτς. Είναι βεβαίως, να κοιτάξουμε τους δικούς μας αλλά γιατί δεν έχουμε, άμα έχουμε μια πρόταση δική μας, γιατί δεν τη θέτουμε στο τραπέζι. Η πραγματικότητα είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Φυσικά δεν είμαστε τυφλοί σε σχέση με αυτά που γίνονται σε ένα διεθνές πλαίσιο. Αλλά οι δικές μας ε, προτεραιότητες είναι αυτή τη στιγμή τα φθοριο, φθοριούχα αέρια και οι εκπομπές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέποντας τι θα γίνει θα δούμε ποιες είναι και οι σωστές πολιτικές επιλογές σχετικά. Κύριο Σκυλακάκης. Θα ήθελα και εγώ να καταγραφεί το εξή: Όταν έχουμε μία επιλογή που κοστίζει 4 ή 5 σεντ τον τόνο ή 20 σεντ τον τόνο και πληρώνουμε 14 θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη ε, φροντίδα και μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και να κρυβόμαστε πίσω από τις διαδικασίες. Η Κομισιόν έχει δράσει για τους HFC-23 με μεγάλη ταχύτητα και με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποτελεσματικότητος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας και τις πρωτοβουλίες μας γιατί αυτό δεν αφορά μονάχα την σωτηρία του πλανήτη, αλλά και την μείωση του κόστους. Ε, εντάξει, λέω ο πρόεδρος, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον καθηγητή Τσέλκε που ήλθε στην Επιτροπή μας. Σίγουρα θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση και η ανάλυση σας θα δοθεί και στα άλλα μέλη της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου και θα παρακολουθήσουμε και την πρόοδο η οποία λαμβάνει η χώρα για τη μείωση αυτών των εκπομπών και έτσι να συμβάλλουμε στην προστασία του κλίματος. Σας ευχαριστούμε καθηγητά Ζέλκε για τις πληροφορίες που μας δώσατε και θα μείνουμε σε επαφή. Σας ευχόμαστε κάθε τύχη. Σημείο 23 τώρα της Μεσσίας διάταξης. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. συγγνώμη, 23. Όχι, έχουμε το 31 όμως προηγουμένως. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. Η νομοθεσία λέει στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν είναι παρούσα για το ερώτημα του Ρίχαρτ Ζέιμπερ για το ΡΙΤΣ. Οπότε δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ερώτημα Ζέιμπερ για να απαντηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι η επικεφαλής των χημικών ουσιών και νανοηλικών. Ο κύριος Ζέιμπερ έθεσε τρεις ερωτήσεις, ε, προσπαθήσω να τις απαντήσω, όχι σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Πρώτα απ' όλα για το τι γίνεται για την εφαρμογή του REACH, ε, γι' αυτό μπορώ να μιλάω με τις ώρες, αλλά να τονίσω έτσι λίγα βασικά ε, σημεία. Πρώτα απ' όλα πέρασε επιτυχώς η πρώτη προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου 2010 υπήρχαν 24.500 ε, ε, και 500 περίπου ε, καταγραφές στην υπηρεσία και έχει τελειώσει ο έλεγχος πληρότητας και βρήκαμε πως 20.750 φάκελοι ήταν πλήρης οπότε 4.500 περίπου φάκελοι θα είναι περισσότερες πληροφορίες. Η προθεσμία αυτή βεβαίως ήταν το σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του κανονισμού, αλλά βεβαίως ε, είναι και η αρχή μιας διαδικασίας, γιατί υπάρχουν άλλες δύο προθεσμίες. Μία είναι και όλα στο 2013 και μία το 2018 για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται χαμηλότερους όγκους. Και άρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δούμε τα μαθήματα από την πρώτη φάση καταγραφής για να γίνει πιο ομαλή διαδικασία μετά. Μετά, η ίδια η καταγραφή είναι ένα βασικό στοιχείο του Ρίτς, αλλά ε, όπως ξέρετε, όπως λέει και η λέξη, υπάρχει αξιολόγηση και περιορισμός τελικά για να ολοκληρωθεί το σύστημα. Όσον αφορά την αξιολόγηση υπάρχουν δύο τύποι, έχουμε τον λεγόμενο φάκελο και την αξιολόγηση ουσίας. Οι αξιολογήσει φακέλου γίνονται από την υπηρεσία, σημαίνει πως η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των φακέλων σε σχέση με τις απαιτήσει που ορίζει το REACH. Αυτή έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Να σας δώσω μια ιδέα. Το 2010 151 φάκελοι εξετάστηκαν, 36% από αυτούς εγκρίθηκαν και οι υπόλοιπες περιπτώσεις είτε βγήκε απόφαση είτε μια επιστολή ε, παρατήρησης, δηλαδή που ουσιαστικά ζητάει περισσότερες πληροφορίες. Ε, δεν είναι και πολύ σπουδαία τα αποτελέσματα, αλλά ε, βεβαίως πρόκειται για την πρώτη καταγραφή, οπότε όλοι μαθαίνουν. Και δεν σημαίνει πως έτσι θα πάνε τα πράγματα και στο μέλλον. Αξιολόγηση ουσιών. Στο ρίτσι γίνεται από την υπηρεσία συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και το γίνεται για να μην υπάρχουν υποψίες βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας ζητώντα πληροφορίε από τη βιομηχανία. Τώρα συλλέγουμε ουσίε και μπαίνουν σε ένα σχέδιο δράσης τη κοινότητα που θα αποτελέσει τη βάση της δουλειά μα και το σχέδιο αυτό δράσης θα υιοθετηθεί το 2012. Όσον αφορά το σύστημα διοδότησης, η Κομισιόν πρόσφατα υιοθέτησε μια απόφαση για να συμπεριλάβει τι πρώτε έξι χημικέ ουσίε στον κατάλογο των ουσιών που θα χρειαστούν αδειοδότηση και αναμένουμε βέβαια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών μια απόφαση για να συμπεριληφθούν άλλες 8 ουσίες ε, από τον κατάλογο των υποψηφίων. Συνολικά ο λεγόμενος κατάλογος των υποψηφίων τώρα έχει τα 46 ουσίες. Όπως ξέρετε η Κομισιόν δεσμεύτηκε πέρσι να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για ένα στόχο να συμπεριληφθούν άλλες 90 ουσίες μέχρι το 2012 και μετά να δούμε όλες τις ε, σχετικές ε, ήδη γνωστές σήμερα ουσίες ε, που θα συμπεριληφθούν μέχρι το 2020, οπότε έχουμε δουλειά μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε από την υπηρεσία για να συμπεριληφθούν άλλες 7 ουσίες και θα έχουμε τους επόμενους γύρους διαβουλεύσεων τον Αύγουστο όσον αφορά τους περιορισμούς. Η Κομισιόν ε, πρότεινε δύο περιορισμούς βασίζονται στις διαδικασίες αξιολόγηση κινδύνου που έγιναν με βάση την προηγούμενη νομοθεσία του ΡΙΤΣ και αφορούν ε, κάδμιο και κουιλαμάιτ αυτέ τι ουσίε. και βεβαίω εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοπεύουμε σύντομα να υποβάλουμε μια τροποποίηση στο παράρτημα 17 που θα συμπεριλάβει τον περιορισμό για την πόλη στο γενικό κοινό ουσιών οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ε. και βλάπτουν το αναπαραγωγικό σύστημα. Οπότε ε, αυτά όσον αφορά την εφαρμογή του ρίτς. Μετά ο κύριος Ζέμπερ ρώτησε το εάν ε, θα, θα χρειαστεί αναθεώρηση του κανονισμού εδώ πέρα να επισημάνω πως ο κανονισμός ο ίδιος προβλέπει αναθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν και να έχουμε βεβαίως τη βάση απόφασης για το εάν θα προτείνουμε αναθεώρηση. Αναμένουμε λοιπόν 1η Ιουνίου 2012 μία αναθεώρηση που θα γίνει από την υπηρεσία. Η λεγόμενη αναθεώρηση χαμηλών χαμηλού τονάζ για τις ουσίες μεταξύ ενός και 10 και μετά βεβαίως υπάρχει και η αναθεώρηση πεδίου εφαρμογής που κοιτάει κενά ή αλληλεπιδράσεις με άλλες νομοθεσίες με άλλα νομοθετήματα γιατί μιλάμε για 160 νομοθετήματα Βεβαίω με την ίδια προθεσμία Ιούνιο 2012 θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση για την εμπειρία μας από τη λειτουργία του ΡΙΤΣ, το δε ποσό που έχει η Κομισιόν να διανύμει για δοκιμές εναλλακτικό, για ε, εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών και βεβαίως αναμένουμε και την έκθεση του ΕΚΑ για τις δικές τους εμπειρίες. Αυτά προβλέπονται ήδη στην ομοθεσία. Αποφασίσαμε όμως να γίνει μια γενικότερη αναθεώρηση το 2012 και άρα δεν θα απαντήσουμε μόνο σε αυτές τις αναθεωρήσεις ε, και τις εκθέσεις, αλλά θα έχουμε έκθεση για τα πρώτα μαθήματα που αντλήθηκαν και για όσον αφορά το κόστος και το διοικητικό άκτος που προέκυψε από το Ρίτς, αλλά βεβαίως και την καινοτομία. Σκοπεύουμε όλα αυτά να βγουν ως πακέτο 1η Ιουνίου 2012 και ε, για την διαδικασία αυτή ξεκινήσαμε πολλές θεματικές μελέτες για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Και όταν θα έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες θα κάτσουμε να τις αναλύσουμε για να δούμε αν χρειάζεται μία αναθεώρηση και βεβαίως τότε θα πρέπει ε, να σκεφτούμε πως έχουμε πλησιάσει, θα έχουμε πλησιάσει τότε τη δεύτερη προθεσμία καταγραφής και να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος πιθανής αναθεώρησης τότε. Τέλος, για να τελειώσω. Ε, ένα ερώτημα για το αν χρειάζεται να επεκταθεί το Ρίντ. Αυτό μας το ρωτάνε συχνά. Υπάρχουν δύο ζητήματα που συχνά αναφέρονται. Το ένα είναι νανοηλικά και το άλλο τα λεγόμενα αποτελέσματα των χημικών κοκτέιλ. Για τα νοηλικά το Κοινοβούλιο ζήτησε να ξαναδούμε την ε, νομοθεσία την σχετική και ε, να κάνουμε μια έκθεση. Αυτό το κάνουμε ήδη και βεβαίως ε, ε είπατε πως ήταν κάπως έτσι επιφανειακή αυτή και θέλετε κάτι πιο πολύ σε βάθος. και πως θα έπρεπε να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να δούμε αν θεωρούμε πως υπάρχει επαρκής διατύπωση του ρίτς για να δούμε τις προκλήσεις των νανοηλικών. Όσον... Σε ό,τι αφορά τα κοκτέιλ όμως, η έκθεση σε πολλαπλά κοκτέιλ από διάφορες προελεύσεις είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φορές δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε με μόνο με χημικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική έκθεση σε κοκτέιλ. Εδώ το Συμβούλιο μας ζήτησε το, Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο του 2009 να κάνουμε μια μελέτη για να δούμε αν χρειάζεται δράση και αν πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη με δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αυτά και τώρα προσπαθούμε να δώσουμε αυτή την έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι το 2012, ώστε να έχουμε μια περαιτέρω σκέψη, δυνατότητα σκέψης σε σχέση με τα κοκτέιλ και την ανάγκη επέκτασης του ρίτς για να καλύψει όλα αυτά τα κοκτέιλ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζέμπερ, θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα επίσης σαν μέλος της Επιτροπής. Όταν εγκρίναμε το REACH, μία από τις εκτιμήσεις που είχαμε ακούσει τότε από την Κομισιόν για τον ε, αντίκτυπο στην ε, χημική βιομηχανία ήταν θα οδηγούσε σε συμπερίληψη στον κατάλογο αυτό 2 με 4.000 επικινδύνων ουσιών στα επόμενα χρόνια. Αλλά τα νούμερα που δίνεται τώρα μαζί με τα κοκτέιλ, ακόμα και αν δεν ξέρουμε πόσες ουσίες δεν συμπεριλαμβάνονται, γιατί πολλές από αυτές είναι ακόμα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ε, αξιολογήσετε αυτές τις εκτιμήσεις που έχετε για τις ουσίες αυτές ή αν έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσες ουσίες θα βγουν πια από την αγορά ως επικίνδυνες μετά από αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας δώσω άλλες πληροφορίες πιο επακριβείς για το θέμα αυτό. Αλλά βρήκαμε και έχετε απόλυτα δίκαια σε αυτά τα σημεία ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ του αριθμού των ουσιών που περιμέναμε να καταγραφούν με την πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την ε, καταγραφή τους και του αριθμού των ουσιών που τελικά παρουσιάστηκαν. Ξεκινήσαμε λοιπόν να λειτουργούμε τον φορέα του και είδαμε ότι υπήρξαν και ορισμένοι λόγοι που μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας. Κάποιες <clears throat> εταιρείε βρήκανε ότι οι ουσίες που αυτοί νομίζαν ότι ήταν διαφορετικές και ήταν στην αγορά με διαφορετικά ονόματα τελικά ήταν η μία και η αυτή ουσία. Και ο δεύτερος λόγος, ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη από μας επαρκώς, ήταν ότι οι μέθοδοι ε, υπολογισμού για, τα, για τις υποκατάστατες ουσίες βάσει της παλιάς νομοθεσίας και της νέας νομοθεσίας ήταν διαφορετική. Στην παλιά νομοθεσία υπολογίζαμε ότι περνούσε το όριο των χιλίων τόνων αν για 15 χρόνια η παραγωγή ήταν πάνω από, ένα, από χιλιούς τόνους το χρόνο. Το REACH όμως είναι νομοθεσία, κοιτάζει μονάχα τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την καταταληκτική προθεσμία καταγραφή και κοιτάζει το μεσόωρο και αν είναι πάνω από χίλιου τόνους αυτή η παραγωγή, τότε η ουσία αυτή εμπίπτει στον κανονισμό του ΡΙΤΣ. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ διακυμάνσει και στο θέμα αυτό και επομένω μαζί με τη χημική βιομηχανία καταλήξαμε στο γεγονό ότι είναι πολύ δυναμική η αγορά χημικών προϊόντων. Έχουμε ουσίες και ουσίες οι οποίες έρχονται μερικές φορές στην αγορά για λίγα χρόνια και μετά εξαφανίζονται και αυτή η εξαφάνισή τους μπορεί να οφείλεται σε εμπορικούς λόγους ή για το γεγονός ότι έχουν έρθει καλύτερες ουσίες οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις προηγούμενες και είναι γεγονός ότι, τουλάχιστον έτσι μας είπε η χημική βιομηχανία, ότι ορισμένες ουσίες έχουν αντικατασταθεί από εναλλακτικές ουσίες που στο παρελθόν δεν είχαν αρκετή αγορά για να υποβάλουν ένα φάκελο καταγραφής στο REACH, αλλά στη συνέχεια μπόρεσαν αυτές να υποβάλουν προτάσεις καταγραφής. Αυτό δείχνει γιατί υπάρχουν διαφορές με τις αρχικές μας προβλέψεις, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα ουσιαστικά αποτελέσματα για τις ουσίες που θα εξέλθουν από την αγορά. Θέλει κάποιος να πει κάτι ακόμα. Όχι. Πάμε στο επόμενο θέμα για την βιοπικιλότητα που έθεσε η κυρία Μπελιέ. Η κυρία Κοντέσου από την Κομισιόν έχει το λόγο. Κύριε Κοντέσου, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Είμαι επικεφαλής της ε, μίας εκ των δύο νομικών ε, μονάδων της ε, DG Περιβάλλον. Όσον αφορά τα θέματα βιοποικιλότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει φιλόδοξους στόχους ώστε να περιορίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέχρι το 2020 και να τα αποκαταστήσει όσο Όσο γίνεται η πλήρης εφαρμογή των δικτύων ε, για τα πτηνά αλλά και για τα οικοσυστήματα, ιδίως η εφαρμογή του Natura, είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εμείς ε, θα εκθέσουμε τα μέτρα με τα οποία σκοπεύουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Είναι δύσκολη η επίτευξή τους ε, και το αναγνωρίζουμε αυτό. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην οριστικοποίηση του Natura 2000 όπου καλύπτει 26.000 μέρη και περίπου 60% ε, ε, του χερσαίου, της χερσαίας επικράτειας της Ένωσης τώρα πρέπει να επεκταθεί για, στη θάλασσα ιδιαίτερα για το θαλάσσιο περιβάλλον και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και εξακολουθούμε να προβαίνουμε σε νομικές ενέργειες όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις ε, διατάξεις κλειδιά της οδηγίας ε, Natura. Στόχο είναι η σωστή διαχείριση και αποκατάσταση των ε, χώρων, ο ορισμό ειδικών περιοχών ε, προστασία και συντήρηση και είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση των περιοχών αυτών και η Κομισιόν θεωρεί πω αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω τη ανάπτυξη ε, προγραμμάτων διαχείριση ή αντίστοιχων μέσων για όλου του χώρου Natura 2000 καθώ και έγκαιρη εφαρμογή. Εμεί προωθούμε εμπειρογνωμοσύνη και ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών με προτεραιότητα την ιεράρχηση των ενεργειών, καθώς και προώθηση του στρατηγικού συντονισμού για τις, τη διαχείριση των ενεργειών διαχείρισης και αποκατάστασης. Φυσικά όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση και τα δημοσιονομικά μέσα τα απαραίτητα για την στήριξη του Natura 2000. Η Κομισιόν θα εκδώσει ανακοινωθέν για τη χρηματοδότηση του Natura 2000 φέτος και με τη βάση, επί τη βάση πληροφοριών που έχουν δώσει τα κράτη-μέλη θα ε, περιλαμβάνει εκτιμήσεις ε, για το κόστος του Natura 2000 και θα αποκομίζει διδάγμα ε, από την μέχρι το δεφαρμογή του προγράμματος με στόχο την βελτίωση Τη χρηματοδότηση του Natura 2000 σύμφωνα με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικέ. Η επίτευξη μεγαλύτερη υποστήριξη για την χρηματοδότηση του Natura 2000 υπό τις ε, σημερινές συνθήκες ε, οικονομικής ε, κρίσης είναι μεγάλη πρόκληση για την ώρα. Γι' αυτό και η Κομισιόν υπογραμμίζει τα ωφέλη που έχουμε να κερδίσουμε από τη σωστή διαχείριση του δικτύου και την προώθηση πιο στρατηγικής προσέγγισης προς την χρηματοδότηση του Natura 2000 για την επόμενη οικονομική περίοδο. Τέλος, η Κομισιόν θα συνεχίσει να προωθεί καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών του Natura για τις ε, γέες και τους χώρους ε, Natura 2000 σύμφωνα με τις διατάξεις ε, του άρθρου 6 το οδηγίας περί οικοσυστημάτων. Εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε ενεργά με τομείς κλειδιά και πρόσφατα Έχουμε εκδώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις εξορρυκτικές βιομηχανίες της βιομηχανίες αιωλικής ενέργειας και επίσης σκοπεύουμε να εκδώσουμε κατευθύντες γραμμές για άλλους τομείς κλειδιά όπως τα ποτάμια, οι πλωτές οδοί και οι δατοκαλλιέργειες. Ωστόσο υπάρχει σαφής ρήξη, όπου μάλλον υπάρχει σαφής παραβίαση των, των, των οδηγιών, θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και ο αριθμός των περιπτώσεων που αφορούν παραβίαση των οδηγιών πτηνών και των οδηγιών για τα οικοσυστήματα είναι ένας από τους ψηλότερους στην, ε, δική μας Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ερώτηση? Then we move on Όχι. Αυτές ευχαριστούμε. Και προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη ερώτηση έχει τεθεί από τον Chris Davis και νομίζω είστε εσείς ο ίδιος υπεύθυνο γιατί είναι, αφορά την οδηγία για τα οικοστήματα. Ευχαριστώ. Πρόκειται για παραβίαση ε, από πλευράς Βουλγαρίας. Το πρώτο και πιο, έτσι, πιο γενικό που έχω να πω, η απόφαση για το εάν συγκεκριμένες αποφάσεις θα πάνε από την ε, πρώτη επιστολή σε αιτιολογημένη ε, γνωμοδότηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ε, την επικοινωνία με το κράτος μέλος. Εδώ πέρα είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες από πλευράς Βουλγαρίας και την ανάγκη ανάλυσης νέων πληροφοριών. Όπως είπα, ο διάλογος συνεχίζεται με τις βουλγαρικές αρχές και τις αρχές κομισιών για τις περιοχές εκείνες που είναι υπό την οδηγία των βιοτόπων πτηνών. Πρέπει να πω πως πρόσφατα η βουλγαρική κυβέρνηση έλαβε απόφαση την λεγόμενη 811 ε, του 2010 για το κομμάτι Εσίας για το δίκτυο Natura 2000 στη Βουλγαρία και έχουμε τρεις νέους τόπους και σε άλλα 25 σημεία έχουμε επέκταση του δικτύου και σε ένα μείωση. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης έχουμε 47.000 εκτάρια συνολικά ή 0,4% της επικράτειας της Βουλγαρίας που θα προσθεθεί στο Natura 2000. Κάτι το οποίο ε, καλύπτεται ήδη ε, καλύπτει ήδη το 34% της βουλγαρικής επικράτειας, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ένωση. Αυτά για τη Βουλγαρία όσον αφορά τώρα τον ορισμό της Χερσονήσου Καλιάκα συνεχίζεται η Κομισιόν αναλύει πολλές αντικρουόμενες τεχνικές πληροφορίες που έστειλαν οι παραπονούμενοι και οι βουλγαρικές αρχές ε, όσον αφορά την Χερσόνησο Καλιάκρα για να διασφαλίσουμε πως ε, οι απαιτήσει προστασίας των πτηνών ε, θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ναι. Εγώ μίλησα με την Κομισιόν το μεσημέρι, με τον κύριο Επίτροπο, και είπε ότι η Σλοβενία έχει 27% του εδάφους που καλύπτεται από το, τις περιοχές Natura 2000, οπότε η Βούλγαροι είναι δεύτερη και όχι πρώτη. Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό αυτό, αλλά τι σημασία έχει πόσο μέρος της ε, χερσαίας επικράτειας μιας χώρας καλύπτεται από έδαφος Natura 2000 εάν οι απαιτήσει δεν εκπληρούνται. Αυτό είναι μια δοκιμασία λοιπόν για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές ομάδες οικολόγων θεωρούν ότι αυτό είναι κομβικό για να καταλάβουμε αν η Κομισιόν θα λάβει πράγματι μέτρα κατά της βουλγαρικής κυβέρνησης. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες, είναι πολύ δάπανο. Αλλά και πιστεύω τα στοιχεία σας το υποστηρίζουν, ότι υπήρξε μια σαφής παραβίαση των κανόνων της Natura 2000. Έχει η Κομισιόν λοιπόν τα κότσια να φέρει τη Βουλγαρία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή θα καθυστερήσετε και θα χρονοτριβήσετε και θα διστάζετε για πολλά χρόνια ελπίζοντας ότι οι διαμαρτυρώμενοι και οι διαδηλωτές για τα θέματα αυτά θα σταματήσουν και θα βαρεθούν. Έχετε τα κότσια λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε, έχουμε, θα είχαμε κανονικά τα κόσια για να προχωρήσουμε σε αυτό, αλλά όπως ξέρετε το βάρος αποδείξεως είναι σε εμά, πάνω σε εμά την Κομισιόν. Αν πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να παρουσιάσουμε ισχυρή επιχειρηματολογία. Και εδώ σας λέω ότι έχουμε πληροφορίες όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι έχουν καταθέσει την αναφορά διαμαρτυρίας, αλλά και από τη βουλγαρική κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν αυτές τις τις αντιπαραθυθέμενες απόψεις να τις αναλύσουμε. Δεν προσπαθούμε να καθυστερήσουμε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για μας οι διατάξεις της οδηγίας για την Natura 2000 να την χάνουν πλήρους σεβασμού ακόμα και από τους Βούλγαρους. Είναι θέμα ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών από την Κομισιόν. Αλλά σα λέω και πάλι σε τέτοιου είδου περιπτώσει και σε τέτοιε υποθέσει τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα διότι εμπλέκονται και ζητήματα χρηματοδότηση. Εμεί δεν προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο για τη Βουλγαρία, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση ώστε αυτέ οι διατάξει να τηρούνται πλήρω και στην Χερσόνησο Καλιάκ. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω ότι δεν καθυστερώ τα άλλα μέλη τη επιτροπή λέει ο κ. Ντέιβι. Επιτρέψτε μου όμως να επανέλθω. Από ό,τι καταλαβαίνω, η διαδικασία επί παραβάση αφορά την λαθασμένη, το λαθασμένο χαρακτηρισμό και τη βλάβη προς το περιβάλλον της χερσόνησης της Καριάκας και αυτό χρονίζει εδώ και τρία χρόνια. Προφανώς πρέπει να ζυγίσετε τα στοιχεία. Αλλά τι χρειάζεται να γίνει μέσα σε τρία χρόνια. Υπάρχει μια περίπτωση, κάποιος πηγαίνει και ελέγχει αυτή την κατάσταση. Αν ήταν τοποθεσία Natura 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγώ νομίζω ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα μπορούσα να σας πω αν υπάρχει ή όχι παραβίαση. Μπορεί η κυβέρνηση να χρειαζόταν δύο μήνες για να απαντήσει στις επιστολές. Πείτε ότι χρειάζονται έξι μήνες αλληλογραφίες. Γιατί όμως τρία χρόνια. Μετά θα είναι άλλα τρία χρόνια και μετά άλλα τρία χρόνια. Μήπως θέλετε μια καταληκτική ημερομηνία για να φέρετε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όχι. Όπως είπα, ο στόχος μας είναι να λυθεί το πρόβλημα και να εφαρμοστούν οι λόγω διατάξεις στη Βουλγαρία όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολλά τα σημεία και αιωλικές εγκαταστάσεις και χρειαζόμαστε πολλές πληροφορίες και από τη Βουλγαρία. Είχαμε πολλές ανταλλαγές, συναντήσεις. Οι τελευταίες πληροφορίες από πλευράς Βουλγαρίας ε, μας τάλησαν το Δεκέμβριο και τις μελετάμε. Έχουμε και άλλη μια συνάντηση στη Βουλγαρία και θα πάμε και επί τόπου, τον Απρίλιο, να δούμε τι συμβαίνει προφανώς όλες οι πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, Κοιτάξτε, η κατάσταση αλλάζει και πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε μια κατάσταση η οποία είναι ενισχυτική και είναι παραβίαση και συζητώντας με τους παραπονούμενους και τις αρμόδιες αρχές να αλλάξει η κατάσταση και πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Οπότε τα πράγματα τρέχουν. Υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που δουλεύουν μόνο και παίρνουν λεφτά μόνο εάν κερδίσουν. Δηλαδή νομίζω πως έχει αρκετά στοιχεία να, να τα δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους και θα βγάλουν λεφτά από τη Βουλγαρία και μοιραστείτε τα λεφτά. Ε, δεν βάλτε τα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γιατί εμένα μου φαίνεται πως συνεχίζεται, πάπυρον Και ε, τίποτα, ε, χρονοτριβείτε. Πρέπει να βάλετε μία προθεσμία και να μας πείτε, να μας δώσετε μία εγγύηση, εν πάση περιπτώσει, ότι θα ξανάρθετε σε τρεις μήνες να μας δώσετε μία απάντηση. Μία πρόοδο όμως. Να σας δώσω έξι μήνες. Μπορείτε σε έξι μήνες να έρθετε να μας πείτε αν έχει επιληθεί το θέμα ή αν έχει γίνει το επόμενο νομικό βήμα και έχει εκδώσει δηλαδή αιτιολογημένη γνώμη. Ναι, ευχαριστώ. Να επανέλθουμε με όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε αυτή τη στιγμή πως θα κάνουμε το επόμενο βήμα ή θα κλείσει η υπόθεση. Αυτό εξαρτάται από την ανάλυση, από πολλούς παράγοντες. Όπως είπα είναι περίπλοκη η υπόθεση. Για να πάμε ενώπιον του ΔΕΚ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Με συγχωρείτε που διαφωνώ εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να το δώσουμε σε ένα δικηγόρο για να πηγαίνει στο δικαστήριο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω άλλη μία ερώτηση και θα ζητήσω την Κομισιό να επανέλθει. Απλά να πω, εντάξει, το ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι και την Κομισιόν και, και τη βουλγαρική κυβέρνηση. Αλλά εάν είναι να δούμε την προστασία των ε, Natura 2000, ε, κάποια στιγμή θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί ο νόμος. Συμφωνώ. Και πρέπει να πω πως είναι θετικό το ότι έχουμε τώρα την ε, ε, δέσμευση της Κομισιόν πως θα επανέλθει σε 6 μήνες. Λοιπόν, επόμενο θέμα επικίνδυνα απόβλητα στους βάλτους του Χουέλβα από την Σάτου Χάση. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα, το πρώτο ερώτημα αφορά και αιτιολογημένη γνώμη. Σε αυτή την περίπτωση καταφέραμε να εκδώσουμε μια αιτιολογημένη γνώμη εις βάρο της Ισπανίας. Πέρσι, το Μάρτιο για την κατάσταση στη Χουέλβα όπου η εταιρεία Φερτιμπέρια έριξε 2,5 εκατομμύρια τόνους μαδρανών υλικών σε ένα βάλτο. Παραβιάστηκαν αρκετές σημαντικές οδηγίες ε, περί αποβλήτων, όσον αφορά βιομηχανικά απόβλητα, ε, περιβάλτων, οδηγία IPPC δηλαδή η άδεια που δόθηκε στην εταιρεία δεν συμπεριλάμβανε όλα τα μέτρα για υψηλό βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, οδηγία χιτά, για το ότι δηλαδή η άδεια της Φερτιμπέρια εκλήρωνε τους απαραίτητους όρους για το απαραίτητο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ισπανία λοιπόν ανέφερε κάποια μέτρα τα οποία ελήθησαν. Δηλαδή αυτό ζητάμε εμείς ένα σχέδιο μέτρων. Μίλησε για αξιολόγηση επιστημονική και σχέδια αναζωογόνησης περιοχής και τι θα γίνει με την κατάσταση. Οπότε υπάρχουν πολλά θετικά βήματα με βάση αυτό το σχέδιο δράσης ε, και ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι σε εκτέλεση μιας εθνικής απόφασης εθνικού δικαστηρίου η Ισπανία ε, προχώρησε στην ε, απομάκρυνση των υλικών αυτών όσον αφορά τη χημική ανάλυση του φωσφορικού γύψου και σύμφωνα με τις αρχές δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με την ε, υφιστάμενη νομοθεσία. Τα ύδατα γύρω από τα απόβλητα όμως θα πρέπει να ε, καθαριστούν στη Λιμνοθάλασσα και μετά αναμένεται να μειωθεί η ρήπανση σε ε, τρεπτά επίπεδα. Ο ραδιολογικός κίνδυνος θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένος η ανάλυση της χημικής φύσης ε, της ουσίας που έπεσε στις ζώνες 1 και 4 συνεχίζεται και η Ισπανία θα μας πει το αποτέλεσμα στην τρίτη έκθεση πρόοδου. Επίσης είπαμε στην Ισπανία πως θα πρέπει να αναφέρει κάθε 3-4 μήνες. Νομίζω έδωσαν την τελευταία έκθεση το Φεβρουάριο. Η Ισπανία επίσης ξεκίνησε τη διαδικασία αλλαγής ε, των αδειών IPPC περί υπογείων υδάτων, ε, διάθεσης αποβλήτων ε, και επανόρθωσης και έχει δει τις τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές της απομάκρυνσης του υλικού. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή λοιπόν θα πρέπει να χτιστούν 10 χώματερες, 10 νέες χώματερες και οι διαφορετικές δράσεις που σχετίζονται με αυτό όσον αφορά δηλαδή την κατασκευή και χρήση των χωματερών θα επεκταθούν σε 7 χρόνια και μιλάμε για α, μισό δισεκατομμύριο ευρώ, οπότε δεν το θεωρούν εφικτό οι αρχές και επέλεξαν μια αποκατάσταση επιτόπου. Ε, ένα πιλωτικό έργο έγινε το 2010. Η αποκατάσταση επιτόπου και βεβαίως ε, το κλείσιμο της παράνομης χωματερής μέχρι το 2015 το αργότερο όταν θα πρέπει να έχει επιληθεί η κατάσταση. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε πώς η Ισπανία δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με, όλους, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να βρει μια συμπεφωνημένη λύση και να εξηγήσει τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν στην συνέχεια των συμπερασμάτων ε, της ε, αποστολής διερευνητική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σα είπα, η Ισπανία μας λέει τα της προόδου και αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή το τέλος του 2015. Η Κομισιόν επίσης θα ήθελε να τονίσει πως ε, ανάλογο παράπονο έτοιμα ε, αντιμετωπίστηκε για την Επιτροπή Αναφορών ε, πέρσι. Ε, θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα συμπληρωματικό. Όχι, περνάμε στο ερώτημα που έχει να κάνει με τις κυρίας Χατουχάση για τις ε, ευρωπαϊκές ε, επιθεωρήσεις περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο, Κοσμός της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του περιβαλλοντικού, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη και είναι απαραίτητες, ωστόσο θα πρέπει να αναλυθούν νέες δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, αξίζει να τονίσει κανείς ότι το νομικό πλαίσιο, το κοινοτικό για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και αποτελείται τώρα από την σύσταση του 2001 που προβλέπει τα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρίες στα κράτη-μέλη καθώς και ορισμένες διατάξεις για τις τομεακές περιβαλλοντικές ε, νομοθεσίες τομεακή προσέγγιση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης θα επέτρεπε την προσαρμογή των κριτηρίων επιθεώρησης ε, στην συγκεκριμένη φύση και τους κινδύνους που καλύπτονται. Η Κομισιόν ξεκίνησε την εισαγωγή ειδικών δεσμευτικών ε, ε, απαιτήσεων για τις επιθεωρήσεις σε διάφορες περιβαλλοντικές νομοθεσίες και περιλαμβάνονται δεσμευτικά στην Οδηγία σε ΒΕΖΟ 2 και στην Οδηγία για την συλλογή και αποθήκευση του άνθρακα, την οδηγία για την προστασία των, ε, των ζώων εργαστηρίου, καθώς και την ε, οδηγία για τον έλεγχο των εκπομπών. Ένα σημαντικό επίσης σημείο συνεργασίας ε, με τους εθνικούς επιθεωρητές είναι αυτό που έχει στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας με τις επιθεωρήσεις των κρατών μελών και στόχο έχει την προώθηση και τον συντονισμό. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει πριν από κάποια χρόνια το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εφαρμογή και την Επιβολή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, το ΙΜΠΕΛ. Έχουμε διάφορες δράσεις. Έχουμε αυτές οι επιθεωρήσεις αντιπροσωπεύονται και σε κοινοτικό επίπεδο όπως ε, για παράδειγμα τον περασμένο Νοέμβριο έγινε μια επιθεώρηση για να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο την το επερχόμενο ειδικό καθεστώς ελέγχου στον τομέα της πρόληψης ε, της βιομηχανικής ρήπασης. Το ΙΜΠΕΛ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα των Κομισιόν για το μέλλον. Ωστόσο, παρόλα αυτά, παρόλα από τους ελέγχους, υπάρχει και τομεακή νομοθεσία και συστάσεις για συνεργασία με τους εθνικούς ελεγκτές, όμως η ποιότητα και το επίπεδο ελέγχων αλλά και επιβολής διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Διάφορες εκδηλώσεις έχουν γίνει για την ε, ενημέρωση αλλά και σεμινάρια στα κράτη-μέλη και δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτά ε, συμπεριλαμβάνουν ελλείψεις στις δομές ε, επιβολής της νομοθεσίας, ανεπαρκής έλεγχη, έλλειψη δειγματοληψίας, διώξεις και κυρώσεις. Η κατάσταση αυτή φυσικά δεν είναι διόλου ικανοποιητική. Η περιβαλλοντική υγεία και οι στόχοι της νομοθεσίας περί αποβλήτων δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως ε, σε διάφορα δε οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη. Δεν μπορούν να επιτευχθούν ούτε οι εξοικονομήσεις εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς ε, και πλήττεται και, ε, πλήττεται και η ανταγωνιστικότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μέγας προβληματισμός, υπάρχει στην Κομισιόν σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους ώστε να αναθεωρηθεί το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη διάφορες επιλογές πολιτικές, καθώς και την προσέγγιση της Ένωσης προς τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, είτε με ελάχιστα κριτήρια για τις επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη, μετατροπή σε οριζόντια οδηγία, εισαγωγή συγκεκριμένων δεσμευτικών ε, όρων για τις, ε, τους ελέγχους, η ανάπτυξη μέσων ε, κατευθυντηρίων γραμμών για τις επιθεωρήσεις είναι κάποιες από αυτές τις επιλογές που εξετάζουμε. Τώρα, από την τομεακή άποψη, η αναδιατύπωση που προτείνεται και η πρόταση για νέο, μια νέα οδηγία για μεγάλους κινδύνους με επικίνδυνες ουσίες θα συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τους ελέγχους. Όμως, από την άποψη της γενικής προσέγγισης, οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος για την, ε, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το περιβαλλοντικό κεκτημένο θα μείνει μέσα στο πλαίσιο της ε, ανακοίνωσης για το περιβάλλον που συζητείται από την Κομισιόν και προτείνεται να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό το μέσο προτείνει τη βελτίωση της εφαρμογής σε κοινοτικό επίπεδο, έτσι ώστε η περιβαλλοντική νομοθεσία να εφαρμόζεται καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. ερώτηση. Παρακαλώ. It's not really so much a question δεύτερη ερώτηση, γιατί νομίζω πως το αίτημα της του Χουάση αναφέρει κάποια σημαντικά πράγματα. Νομίζω λοιπόν πως ε, θα πρέπει να δει μια σωστή απάντηση, γιατί είναι θέμα πολιτικής και όχι παραβίασης. Ο εκπρόσωπος Κομισιόν μίλησε για την σύσταση περί ελάχιστων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Όταν ήρθε αυτή η σύσταση στην Επιτροπή μας, το, πότε ήταν, 99-2000, εμείς είπαμε να γίνει οδηγία καμία οδηγία. Καταλήξαμε σε μια σύσταση. Αλλά είναι κάτι που νομίζω πως η Κομισιόν ε, θα πρέπει να το ξαναδεί. Χρειαζόμαστε ελάχιστες περιβαλλοντικές ε, επιθεωρήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο σχόλιο. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, αλλά επειδή οι βουλευτές απουσιάζουν, θα πρέπει να τα δούμε άλλη ώρα. Άρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής. Ο Chris Davis είναι αρμόδιος, αλλά αν δεν σε πειράζει Chris θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Μπούγκουης που είναι παρόν έχει τον λόγο. Thank you, Mr. Chairman. My name is Julio García Burgués, head of the uh, waste uh, Ονομάζομαι Χούλιο Γαρθία Μπουργκές και είμαι επικεφαλής της ε, μονάδας ε, για τις επιθεωρήσεις στην ε, γάμα δέλτα περιβάλλον. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έκανα τα ίδια με τον συνάδελφο Ιωνέσκου, που είναι επικεφαλής ενός από τα τμήματα για την, ε, τα νομικά τμήματα της ε, DG Περιβάλλον. Καταρχήν θέλουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας ELV για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ε, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις νομικές πτυχές και τα εθνικά πακέτα για συστάσεις. Ναι, ναι. ναι. Η οδηγία αυτή έχει αποδειχτεί επιτυχή σε πολλούς τομείς. Έχει οδηγήσει στην μείωση των εγκαταλελειμμένων ε, αυτοκινήτων, στη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων για τη συγκέντρωση όλων αυτών των ε, αυτοκινήτων ε, καθώς και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει συμβάλει στην, στον οικολογικό σχεδιασμό των αυτοκινήτων ώστε να ανακυκλώνονται παραμένουν ορισμένα ε, προβλήματα εφαρμοστικά. Ήδη έχουμε συζητήσει τα προβλήματα αυτά στην Επιτροπή πέρυσι με την ευκαιρία μιας ε, προφορικής ερώτησης που είχε καταθέσει ο κ. Κρίς Ντέιβις. Τα προβλήματα εφαρμογής ε, διαρκώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα ωφελήθει πλήρως από τις διατάξεις της οδηγίας αυτής και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι πλήρως ικανοποιητική. Υπάρχει η βασική απόκληση ανάμεσα στον αριθμό των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής και το αριθμό πιστοποιητικών απόσυρσης ή καταστροφής που εκδίδουν οι πιστοποιητικών απόσυρσης που εκδίδουν ή καταστροφής που εκδίδουν οι εθνικές αρχές. Αυτό σημαίνει πως διάφορα παλιά αυτοκίνητα δεν αναφέρονται σωστά, δεν καταγράφονται και άρα αγνοείται η τύχη τους. Αυτό το πρόβλημα συνδέεται στενά με την ελλειπή εποπτεία της ε, διαδικασίας ε, καταγραφής στα κρατη και εν μέρη στις εξαγωγές οχημάτων ε, στο τέλος του κύκλου ζωής τους που παρουσιάζονται ως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και εξάγονται εκτός της Ένωσης. Πέρυσι ε, είχαμε στη διάθεσή μας τα στατιστικά στοιχεία του 2008 που έδειξαν ε, βελτίωση στην απόδοση των κρατών μελών. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση των νέων στοιχείων που υπέβαλαν τα κρατη Όμως δυστυχώς η πρώτη ανάλυση που έχει γίνει δείχνει πως η πρόοδος δεν είναι αρκετά γρήγορη. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό παλιών αυτοκινήτων που, αγνοεί, που αγνοούνται που δεν έχουν καταλήξει σε ειδικού χώρου συγκέντρωση αυτών των αυτοκινήτων ή που νόμιμα να έχουν εξαχθεί προ τρίτε χώρε. Έχουμε προβεί σε διάφορα διαβήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Καταρχήν, η Κομισιόν έχει ε, εξετάσει το θέμα λεπτομερώς και έχει ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες κατά ε, για... για παραβίαση της νομοθεσίας έναντι διαφόρων κρατών μελών για μη τήρηση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Εξακολουθούν να εκκρεμούν εννέα ε, υποθέσεις και στις περισσότερες από αυτές το βασικό ζήτημα είναι η μεταγραφή της οδηγίας όσον αφορά την καταγραφή των αυτοκινήτων και των πιστοποιητικών καταστροφής τους. Στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων κακής μεταγραφής των οδηγιών είχαμε διμερείς επαφές με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν ήταν επιτυχής. Για παράδειγμα, στην ΟΒ, Βασίλειο το σύστημα καταγραφής αυτοκινήτων έχει αλλάξει και έχει προσαρμοστεί με τις διατάξεις της οδηγίας ELV. Κατά δεύτερο λόγο, ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα των στατιστικών για τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται με, το, με τη μία ρόδα στον τάφο. Τον Απρίλιο εκδώσαμε κατευθυντήρες γραμμές βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίδουν αναφορές για αυτοκίνητα στις εθνικές αγορές, δίδουν συγκεκριμένα και λεπτομεριακά στοιχεία για τα τεταξινομημένα αυτοκίνητα, για τον αριθμό των αυτοκινήτων τα οποία έχουν εξαχθεί όντας μεταχειρισμένα και για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν τύχει ανακύκλωσης κατά τρόπο ο οποίος είναι εγκεκριμένο. Αυτό θα επιτρέψει την Κομισιόν για πρώτη φορά να μπορεί να έχει στοιχεία αξιόπιστα για τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στο τέλος στο παραπέντε και τα οποία δεν αναφέρονται ως αυτοκίνητα στο τέλος της ζωής τους. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κοιτάζουμε επίση τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε την απόφαση αυτή η οποία καθορίζει την μεθοδολογία για τις αναφορές που να καταδεικνύει έτσι καλύτερα το τι συμβαίνει σε αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία γνωρούνται. Τα αυτοκίνητα αυτά όταν εξάγονται σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασίες για την αντιμετώπιση των αποβλήτων, απορριμμάτων και χούφταλοαυτοκινήτων. Ο στόχος μας είναι να εμποδίσουμε, να παρεμποδίσουμε την εξαγωγή αυτοκινήτων στο τέλος της ζωής τους ως αυτοκίνητα εν και έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις στις κατευθυντήρες γραμμές μας για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Παραλλήλως προετοιμάζουμε και μια νομοθετική πρόταση για να ενισχύσουμε τις ειδικέ προδιαγραφές στα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν με την οδηγία ε, εξαγωγών αποβλήτων και απορριμμάτων. Ελπίζουμε λοιπόν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια μελλοντική μεταρρύθμιση της οδηγίας αυτής στο φως των φώτων πορείας και της εμπειρίας που θα έχει κτηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο της τρέχουσας οδηγίας. Δυστυχώς η ικανότητα παρακολούθησης της εφαρμογής αυτής της οδηγίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένες και γι' αυτό εξετάζουμε τις δυνατότητές μας, μεταξύ των οποίων τη δημιουργία ενός φορέα σκουπιδιών, για να μπορεί να παρακολουθήσει την νομοθεσία περί από, αποβλήτων και σκυβάλων. Πιστεύουμε ότι μια καλύτερη εφαρμογή αυτής της οδηγίας είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε τους στόχους μιας σωστής αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και χαιρετίζουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσουμε ότι η αποτελεσματική αυτή εφαρμογή της οδηγίας θα γίνει μία από τις πρώτες προτεραιότητες των κρατών μελών. Σας ευχαριστούμε. Κρίς, θες να πεις κάτι ακόμα. Ναι, ναι, ναι, θέλω. Μα, κύριε Πρόεδρε, μια ιστορική αναδρομή. Ήταν από τις πρώτες οδηγίες που είχα ασχοληθεί για το θέμα αυτό. Ήμουνα εισηγητής με τον Καρλ Χάιντς ε, Φλόρενς πριν από το 1988, 1998 καλύτερα. Καταρχήν είναι πολύ καλή νομοθεσία αυτή. Είναι μια νομοθεσία που αντιμετώπιζε τα 14, 14 εκατομμύρια έκθετα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό <clears throat> ενθάρρυνε την ε, ανακύκλωσή του, την οικολογική σχεδίαση στα αυτοκίνητα, όπως είπε η Κομισιό. Και επειδή ήταν ευρωπαϊκό μέτρο, εξασφάλισε ότι οι κατασκευαστές δεν μπορούσαν να πούν «Α, θα πάμε σε άλλες χώρες». Τελικά αυτό τους υπευθυνοποίησε. Τους ενοχλούσε πάρα πολύ η έννοια της ευθύνη του παραγωγού, αλλά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά δεν είχαν κανένα πρόβλημα για τους κατασκευαστές. Κανένα πρόβλημα δεν τους δημιούργησε. Ενώ τότε λέγανε πω πω θα μας καταστρέψει την αυτοκινητοβιομηχανία. Λοιπόν, όπως είπε και ο τη Κομισιόν, η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το Τμήμα Πολιτική και Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει παρουσιάσει μια μελέτη για την κατάσταση αυτή και ορισμένε συστάσει και χαίρομαι που η Κομισιόν έχει μελετήσει εντελεχώ τι προτάσει του Κοινοβουλίου. Ένα από τα προβλήματα είναι όπως ελεγχθεί ότι είναι εκατομμύρια αυτοκίνητα που είναι αγνοούμενα. Κάπου έχουν πάει στο εξωτερικό, κάποια όμως όχι. Εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο αγνοείται η διαμονή τους, αγνοείται η τύχη τους. Δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ίσως εξάγονται, λαθρέα. Πολλά όμως από αυτά τα αυτοκίνητα είναι σακαράκες. Δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν είναι καρμανιόλες. Δεν πρέπει να είναι στους δρόμους μας. Και τώρα για τα διάφορα θέματα τα οποία γύρονται. Το πρώτο το οποίο έθεσε η Κομισιόν είναι η ελληματική εφαρμογή από ένα αριθμό κρατών μελών και οι διαφορές στον τρόπο εφαρμογής. Χαίρομαι επίση για την Κομισιόν που με βοήθησε στο Ηνωμένο Βασίλειο να μπορέσω να κλείσω αυτό το παραθυράκι το οποίο υπήρχε το οποίο ακύρωνε ουσιαστικά την νομοθεσία αυτή στη χώρα μου για πολλά χρόνια. Με, την, με τον τρόπο που εφαρμοζόταν η νομοθεσία, ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα κάθε χρόνο τα διαλύαν οι ιδιοκτήτες στον καράζ τους και στην αυλή τους. Εν πάση περιπτώσει το κλείσαμε αυτό το παραθυράκι. Ποια είναι τα προβλήματα τώρα. Πρώτα απ' όλα η κακή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Δεύτερον το γεγονός τα στοιχεία συλλέγονται και κρατούνται με διαφορετικό τρόπο και δεν έχουμε συγκρίσιμε στατιστικέ. Τρίτον, το πρόβλημα της λαθρέας εξαγωγής αυτών των αυτοκινήτων. Τέταρτον, ότι η οδηγία δεν έχει σαν στόχο μόνο την ανακύκλωση, αλλά την καταστροφή των ρήπων. Ότι δηλαδή τα απόβλητα από τα αυτοκίνητα δεν μπαίνουν στα ποτάμια και στις λίμνες. Και επανερχόμαστε στο θέμα των ελαχίστων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε πολλά κράτη-μέλη. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση για τις επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος, αλλά είναι μάλλον πολύ ζωφερή σε ορισμένε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται έλεγχος και δεν ξέρω και τι γίνεται με την παρακολούθηση της ανακύκλωσης και το εάν επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Εκεί όπου έχουμε στοιχεία μάλλον ξέρουμε τα νούμερα, αλλά όπως είπα λείπουν τόσα πολλά αυτοκίνητα που τα στοιχεία δεν, δεν καλύπτουν την κατάσταση. Ένα θέμα είναι το ζήτημα του φόρου και αν οι συστάσεις που κάνουμε λαμβάνονται υπόψη. Καταλαβαίνω πως κάποιες χώρες πληρώνει κανείς τέλη κυκλοφορίας μέχρι να φέρει πιστοποιητικό καταστροφής. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι τρόπος για να διαθέσει σωστά ο ιδιοκτήτης το αυτοκίνητό του και δεν ξέρω αν είναι σχαδευτήριες γραμμές. Δεύτερον, το θέμα, το γενικό, πως προετοιμάζονται κατευθυντήριες γραμμές Σωστό αυτό, κάνετε κάτι συνέδρια για να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να δουν την νομοθεσία, αλλά προσκαλέσατε και εμά. Είπατε, Κοινοβούλιο, αυξήστε την πίεση παρακαλούμε. Εμείς θα το θέλαμε, δηλαδή 10 χρόνια σέρνεται η νομοθεσία, προφανώς καλό θα ήταν να έχουμε μια συμφωνία να αναδιατυπωθεί η νομοθεσία. Αλλά πείτε μας τι να κάνουμε για να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν. Βέβαια, τώρα αυτό που λέω... Ε, πείτε μας δηλαδή πώς να σας ασκήσουμε πίεση είναι λίγο αυτοκτονικό. Μα, σας ζητάμε να μας πουλήσετε το σκηνή που θα σας κρεμάσουμε. Αλλά ή να το κατασκευάσετε κιόλας. Την αγχώνει. Εν πάση περιπτώσει πώς να αυξήσουμε την πίεση. Θα απαντήσετε την ερώτηση. Ναι, και γρήγορα. Ευχαριστούμε για την μελέτη αυτή. Με τους τόσους νόμους που έχουμε για τα απόλυτα στην Ένωση, νομίζω μπορούμε να αξιολογήσουμε πως η οδηγία αυτή είναι η πιο ε, επιτυχής στην εφαρμογή της. Υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, παράνομες ε, μεταφορές ε, σε τρίτα μέρη της αβούρας, σε τρίτα κράτη. Το θέμα είναι αν μπορεί να λυθεί αυτό με την οδηγία. Δεν ξέρω. Επίσης να πω πως έχουμε χρήση βαρέων μετάλλων η οποία καταργήθηκε πρακτικά στην αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της οδηγίας αυτής, εκτός από εκεί που δεν υπάρχει βεβαίως ε, εναλλακτική ε, δηλαδή ο μόλυβδος ε, στα... στις μπαταρίες που δεν μπορεί να αντεκατασταθεί με χρυσό. Αλλά έχουμε βαρέα μέταλλα και σε, σε άλλα σημεία πλέον, πριν της αυτοκινητομηχανίας. Οπότε ζητάω από την Κομισιόν τώρα να, να ξαναδεί αυτό το νόμο για να λύσει προβλήματα εφαρμογής. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Το θέμα είναι το αναγκαίο. Εγώ προσωπικά από τη μελέτη, έτσι που έριξα μια ματιά, θεωρώ πως δεν, δεν ε, χρειάζεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αλλού σοβαρότερα προβλήματα με τα απόβλητα που δεν τα ελέγχουμε. Να πω μόνο τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Οπότε σας ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη. Έχουμε επιτυχή νομοθεσία. Υπάρχουν μικρά προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά τίποτα το σοβαρό. Και για αυτό το οποίο είπε ο Chris Davis. Σε κάποια κράτη-μέλη λειτουργεί πολύ καλά η κατάσταση, σε άλλα κράτη-μέλη όχι τόσο καλά. Ε, τώρα να έχουμε το, το φόρο, το, το να λέμε πως θα επιβληθεί φόρο σαράβαλων να πούμε, αυτό τιμωρεί αυτούς τα, τα κάνουν και καλά. Η Κομισιόν. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε. Πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι η μελέτη για τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους που έχετε εκπονήσει ήταν πολύ χρήσιμη για την Κομισιόν. Κύρια, τα κύρια πορίσματά σας βέβαια δεν κομίζουν γλάφκα ούτε καρμπιρατέρ στην Κομισιόν. Αλλά είναι χρήσιμο πιστεύω να γνωρίσουμε τα συμπεράσματά σας για να μας βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή στην πρωτοβουλία μας για καλύτερη εφαρμογή αυτής της οδηγίας να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για την ύπαρξη παραθυρακίων σε μία οδηγία που αντιμετωπίζει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή αυτής της οδηγίας είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μοναχά για την προστασία του περιβάλλοντος και από την πτυχή αυτή του περιβάλλοντος, αλλά και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους δικούς μας στόχους σε ό,τι αφορά την καλύτερη αποδοτικότητα στην χρήση των πόρων. Υπάρχουν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Νομίζουμε ότι ασκώντας τους θεσμικούς του μειώνες μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα υποβληθεί από την Κομισιόν μια πρόταση η οποία θα ενισχύσει τις υφιστάμενες διατάξεις για την επιθεώρηση το, του κανονισμού για την εξαγωγή αποβλήτων και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα Δευτέρας χειρός. Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για τα αυτοκίνητα που πλησιάζουν το θάνατο. Και σε σχέση με τη δυνατότητα να υπάρξει αναδιατύπωση της οδηγίας για τα αυτοκίνητα στο τέλος της ζωής τους, για μας, προς το παρόν, η προτεραιότης είναι σαφώς η επίτευξη της καλύτερης εφαρμογής της υφιστάμενης οδηγίας. Υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο απόδοσης των κρατών μελών εφαρμόζων την οδηγία αυτή. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε μια πιο ισόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και να παροτρύνουμε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν αποδώσει ιδιαίτερα για να βελτιώσουν του, τους βαθμούς τους. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι κεφαλαιόδες και πιστεύουμε ότι έχουμε επιτύχει και κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη πληροφόρηση προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κατάσταση, με το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη για τα ατυχή αυτά αυτοκίνητα. Υπάρχουν όμως ακόμα χάσματα πληροφόρησης. Πάντως είναι πολύ καλύτερη η εικόνα που έχουμε τώρα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα. Σύντομα. Να απαντήσω στο σχόλιο Κράμερ. Εντάξει, σωστό αυτό. Αν δούμε όλα τα, τα ηλεκτρικά απόβλητα, όλη την νομοθεσία περί αποβλήτων, ε, τίποτα δεν είναι στο 100%. Κάποια απέχουν και πάρα πολύ. Και αυτή η νομοθεσία τα πάει καλύτερα βεβαίως. Αλλά υπάρχει, υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών τεράστιες. Κάποια κάνουν τα πάνε εξαιρετικά, κάποια άλλα όχι τόσο. Όπω λένε και στο management, 10 μέτρα και μια κόβε. Δηλαδή καμιά φορά δεν ξέρουμε τι, τι, μετρά, τι προσπαθούμε να μετρήσουμε. Είμαστε 50% του στόχου, στο 100% του στόχου. Δεν υπάρχει ο στόχο ω απόλυτο αριθμό. Δεν ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα βγαίνουν εκτό κυκλοφορία από τον τελευταίο εγχώριο ιδιοκτήτη σε κάθε χώρα. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θεωρεί πως μπορούμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Ένας συνδυασμός δηλαδή όσων πάνε προς ε, εξαγωγή και σκράπ. Εάν μπορούσαμε δηλαδή ανακράτος μέλος να έχουμε τις διάφορες απαιτήσει για να έχουμε αυτήν την αξιολόγηση θα είχαμε καλύτερη εικόνα για το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία και πού έχουμε αδυναμίες. Η Κομισιόν έχει μία απάντηση. Ε, μόνο να πω πως ε, αυτό ακριβώς είναι ο στόχος μας να έχουμε ε, μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και πάλι ε, δεν είμαστε εκεί, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε αλλά πλησιάζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά για αυτό το θέμα τη ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο επανεξέταση τη κοινοτική στρατηγική για τον Ιδράργυρο. Κύριο Σνάμπελ είναι εδώ από την Κομισιόν, έχει το λόγο. Yes, good afternoon, uh, Mr. Chairman. καλησπέρα σας, είμαι ο Κριστόφ Αλέν από την Κομισιόν. υιοθετήσαμε το Δεκέμβριο πέρσι την ανακοίνωση 2010-273 περί αναθεωρήσεως της κοινοτικής στρατηγικής για τον Ιδράργυρο. Επανεξετάζει τη στρατηγική που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν το 2005 και με βάση την οποία είχε ε, υιοθετήσει ψήφισμα το Κοινοβούλιο και κοίταζε και τις εσωτερικές πολιτικές και την παγκόσμια πτυχή του Ιδραργύρου. Υπ' αυτή την έννοια έπαιξε ένα καινοτόμο ρόλο καθώς η διεθνή συνειδητοποίηση για την ανάληψη δράσης δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Σήμερα, μετά την αναθεώρηση, που κάναμε πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής βλέπουμε πως έχει λάβει χώρα σημαντική πρόοδος. Και οι 20 δράσεις ε, που υπήρχαν σε αυτή τη στρατηγική έχουν είτε εφαρμοστεί είτε είναι σε καλό δρόμο. Να επισημάνω τρία νομοθετήματα που υιοθήθηκαν από το 2005 και αποτελούν τμήμα των επιτευγμάτων μας η οδηγία του 2007 περί περιορισμού ορισμένων ε, εμπορίας συσκευών μετρήσεων με υδραργύρου ε, βγάλε κάποια πράγματα από την αγορά, π.χ. τα θερμόμετρα ε, για οικιακή χρήση. Το 2008 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εθέτησαν τον κανονισμό απαγόρευσης εξαγωγών υδραργύρου και αποθήκευση σιδηραργύρου και αυτό έστειλε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Η απαγόρευση εξαγωγών ετέθη ισχύ πριν από λίγες ημέρες. Τέλος, το 2010, η νέα οδηγία βιομηχανικών εκπομπών ε, υιοθετήθηκε και σύμφωνα με την οδηγία ε, καταλήξαμε στις καλύτερες δυνατές ε, τεχνολογίες οι οποίες πλέον θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον ορισμό τιμών ε, εκπομπών. Τα συμπεράσματα βεβαίως πρέπει να υιοθετηθούν από την Κομισιόν. Θα υιοθετηθούν τομέα που καλύπτεται από την στρατηγική και βεβαίως συμπεριλαμβάνει και ε, τον υδράρχηρο και την ε, βιομηχανία ε, αλκαλίων και τα μεγάλα εργοστάσια καύσης, τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Οπότε η ενίσχυση αυτή τη πτυχή στην νομοθεσία θα αποτελέσει αφορμή μείωση του υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν γύρω στις 20 δράσεις στη στρατηγική αυτή, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες όλων των δράσεων, αλλά θα ήθελα να τονίσω πως υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η δράση της Ένωσης στο διεθνές επίπεδο έπαιξε κέριο ρόλο στην απόφαση που ελήφθη το Φεβρουάριο του 2009 από το ΔΣ του προγράμματος του περιβάλλοντος του ΟΗΕ για να υπάρξει μια διαπραγματευτική επιτροπή για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο το οποίο θα καταστήσει δυνατό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί για την κατάργηση της πρωτογενούς παραγωγής και να ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να σταματήσουν να διαθέτουν στην αγορά τα πλεονάσματά τους. Πού είναι βασικός στόχος ε, της στρατηγικής μας. Είναι ιδιαίτερο θετικό πως η διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να επικεντρώσει προσπάθειε και τους πόρους της στις ε, διαπραγματεύσει αυτές. Η διαδικασία ε, θα ολοκληρωθεί το 2013, αρχέ του 2013. Δράτω με τη να σας ενημερώσω πως ε, η Κομισιόν απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπή σα. Η επιστολή είναι καθοδόν και περιέχει τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων. Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις, όπως είπα, είναι θετικές, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει από την πρόοδο στο εσωτερικό. Να αναφέρω τώρα τρεις σημαντικές δράσεις που συνεχίζονται για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή. Αυτή τη στιγμή, υπό την ηγεσία της Υπηρεσίας Χημικών, αξιολογούμε τις επιλογές για, μελλοντικές, ε, για μελλοντικούς περιορισμούς ε, στην εμπορία συσκευών που περιέχουν υδράργυρο και πλέον μιλάμε για τα πιεσόμετρα δηλαδή. Που και αυτό συμπληρώνει τον προηγούμενο κανονισμό που απαγόρευε τη χρήση εξοπλισμού κατοίκων οικιακού εξοπλισμού. Μια άλλη δράση είναι ο καθορισμός περιβαλλοντικών κριτηρίων για την ασφαλή αποθήκευση υδραργύρου. Σκοπεύουμε να ειδητήσουμε τα κριτήρια πριν από το καλοκαίρι με εφαρμοστική πράξη του κανονισμού του 2005 και τα κριτήρια αυτά καλύψουν την προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου και χρειαζόμαστε περισσότερες, περισσότερη δουλειά για πιθανή αποθήκευση του μόνιμη υπογείως. Τρίτον, εξετάζουμε τώρα τις περιβαλλοντικές πτυχές των σφραγισμάτων που περιέχουν υδράργυρο και συλλέγουμε πληροφορίες για εναλλακτικές για α, τις μπαταρίες τις πολύ μικρές μπαταρίες ε, ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτές είναι οι βασικές χρήσεις που απομένουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος, να τονίσω πως για έναν επίμονο ρήπο που ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις και είναι βιοσυσσωρεύσιμος, η η δράση της Ένωσης δεν θα επιτρέψει από μόνη της να επιτύχουμε τους στόχους μας. Οπότε, ενώ δρόμος στο εσωτερικό, έχει τρομερή σημασία να κινητοποιηθούμε σε διεθνές επίπεδο για να επιτύχουμε μια διεθνή συμφωνία οποία θα είναι όσο δυνατόν πιο φιλόδοξη. Ένα πάρα πολύ σύντομα ερώτημα μονάχα. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Είναι βέβαια τοξικός ο υδράργυρος, θα πρέπει να αποφευθεί η επαφή μαζί του και η Κομισιόν έχει παρουσιάσει πολύ ε, πλήρη στοιχεία για τα προϊόντα αυτά, τα οποία καλύπτονται από νομοθετικές ε, ρυθμίσεις και πρέπει να αποφεύγεται ή απαγορεύεται η χρήση τους όργανα μέτρησης παραγωγής χάρη σε οικιακό επίπεδο έχουν μια πολύ μικρή αγορά. Τα περισσότερα είναι βιοτεχνικής παραγωγής, αναφερθήκατε και στις μπαταρίες, στα σφραγίσματα. Θα ήθελα να γνωρίσω αν η Κομισιόν θέλει να αποαπαγορεύσει στα φωτιστικά τον υδράργυρο, τα οποία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ιδίω σε οικιακό επίπεδο και υπάρχουν επίσης μελέτες που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που προέρχονται από παλιά, παλιάς τεχνολογίες φωτιστικά, όταν παραδείγματος σπάσουν οι λαμπτήρες. Τι έχει να προτείνει η Κομισιόν για τη χρήση του υδραργίου σε φωτιστικές συσκευές. το περιεχόμενο σε επικίνδυνες ουσίες που έχουν αυτές οι λάμπες υπόκειται στην οδηγία για τις επικίνδυνες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Υπήρξε μια συμφωνία για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που οδήγησε στην έγκριση αυτής της μεταρρύθμισης πέρσι. Βάσει αυτής της ε, μορφής της οδηγίας. Το περιεχόμενο σε υδράργυρο σε αυτές τις λάμπες είναι περιορισμένο. Περιορίζεται σε 5 μιλιγραμμάρια και η αρχή της οδηγίας αυτής είναι ότι εάν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις τότε δεν μπορεί να δίδεται εξαίρεση ή περιορίζεται η προσφυγή στην εξαίρεση η οποία θα επέτρεπε τη χρήση υδραργύρου σε τέτοιο εξοπλισμό. Εμείς παρακολουθούμε το περιεχόμενο του υδράργυρου σε αυτές τις ε, λάμπες και έχει ληφθεί, έχει ληφθεί μια απόφαση από την Κομισιόν η οποία θα μειώσει το επιτρεπόμενο επίπεδο παρουσίας σε 3,5 μιλιγκράμμ τον Δεκέμβριο και 2,5 μιλιγκράμμ μετά από ένα χρόνο το Δεκέμβριο του 2012. για τα δυνητικά αποτελέσματα της παρουσίας του υδραργύρου στην ανθρώπινη υγεία. Υπήρξε μια γνωμοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή για τα θέματα αυτά, η οποία αφού ανεδίφισε την επιστημονική βιβλιογραφία, δεν μπόρεσε να καταλήξει σε επίπεδο κινδύνου όταν σπάνε αυτές οι λάμπες, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την έκθεση. Βέβαια, όταν σπάει μια τέτοια λάμπα υδραργύρου σε ένα νοικοκυριό θα πρέπει να παίρνουν ορισμένες προφυλάξεις. Και αυτό γίνεται σε, σε κάποια κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο όμως ενέκρινε πρόσφατα ένα συμπέρασμα σε σχέση με τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για αυτά τα προβλήματα που περιλαμβάνει και μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη αλλά και προς την Κομισιόν να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση του κοινού σε σχέση με θέματα τα οποία άπτονται του Ιδραργίου. Ευχαριστώ, είσαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και προχωρούμε. Η προφορική ερώτηση μεταξύ άλλων από τον κύριο Ποκ για τις ελλείψεις και ανεπάρκειες της σημερινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καρκίνο του ορθού Δίνω το λόγο στην Κομισιόν λοιπόν και ο κύριος Πότση ίσως έχει το δικαίωμα θα θέλει να λάβει το λόγο μετά. Έχει το λόγο πάντως η Κομισιόν. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Στέφαν Στέκ, αντιπροσωπεύω την Γενική Διεύθυνση Υγεία και Καταναλωτή. Επειδή υπάρχουν τρει ερωτήσει και μία ερώτηση αφορά περισσότερο την έρευνα, έχω μαζί μου τη συνάδελφο Μαρία Φιντέλ που θα απαντήσει στην ερώτηση υπαριθμών 2. Εγώ στην 1 και στην 3. Η τρίτη ήταν πότε σκοπεύει η Κομισιόν να δημοσιεύσει τι κατευθύνε γραμμέ για την ανείχνευση του καρκίνου του ορθού και γιατί υπήρξε καθυστέρηση σίγουρα γνωρίζετε, δημοσιεύσαμε την πρώτη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών στι 3 Φεβρουαρίου 2011. Έχουν δημοσιευθεί με καθυστέρηση μεν, αλλά δημοσιεύτηκαν. Και το πεδίο εφαρμογή ε, μπορεί να εξηγεί την καθυστέρηση, γιατί οι κατευθυντήριε γραμμέ ε, αντιπροσωπεύουν την κοινή εργασία 90 εμπειρογνωμόνων από 30 χώρε. Έχουμε 400 ε, σελίδες 450 συστάσεις ε, με 750 παραπομπές σε επιστημονικά άρθρα και μόνο η περιγραφή των ε, αποδείξεων που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν σε τυπωμένη μορφή, είναι ένα έγγραφο χιλίων σελίδων. Και αυτό σας δείχνει ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στο να φτιάξουμε κάτι από κοινού για τα 27 κράτη-μέλη, αντί μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος. Τέλος, θα ήθελα να πω πως είναι σημαντικό να σημειώνουμε επίσης πως οι κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα έχουν συναγραφτεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα για τον Καρκίνο στην Λιόν. Και εμείς δεν θέλαμε να παρέμβουμε στην ε, επιστημονική διαδικασία και γι' αυτό και είχαμε περιορισμένο αντίκτυπο στο χρόνο που χρειαζόταν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και τη συγγραφή των κατευθυντηρίων γραμμών. Και τώρα έρχομαι στην πρώτη ερώτηση για τα πρόσθετα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Κομισιόν για να επιταχύνει την εφαρμογή, τα τα... για να επιταχύνει τα προγράμματα με βάση τον ε, πληθυσμό για την ανείχνευση του καρκίνου του ορθού. Η υψηλή ποιότητα ανείχνευση δίνει την ευκαιρία να λάβει κανείς έγκαιρη ε, θεραπεία η οποία μπορεί να του σώσει τη ζωή. Έχουμε το FOBT που είναι ένα ειδικό αιματολογικό έλεγχο και περιορίζει το, ε, την, την ε, περίπτωση της, ε, της νόσου σε ανθρώπους 50 με 74 χρονών κατά, <coughs> κατά 50%. Οι συστάσεις λοιπόν δείχνουν ότι από τα τρία προτινόμενα, τις τρεις προτινόμενους ε, τρόπους ανείχνευσης, το, η ανείχνευση μέσω κολονοσκόπησης είναι η καλύτερη μέθοδος ε, Αυτά δείχνουν οι επιστημονικές μαρτυρίες. Πρέπει να γίνει λοιπόν επιταχυμένη χρήση αυτών των ελέγχων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία. Η επιβολή τέτοιων προγραμμάτων ανείχνευσης του καρκίνου σε, ολόκληρο το, σε, σε, μια ολόκληρη χώρα οφείλεται, ε, μάλλον ε, μπορεί να πάρει και 10 χρόνια λόγω της ανάγκης μετάφρασης των οδηγιών, της ε, ε, μεγάλης ε, κλίμακας ε, προγραμμάτων που υπάρχουν. Έχουμε τώρα τουλάχιστον τις κατευθυντήριες γραμμές και ιδιαίτερα έχουμε και τη συνεργασία μέσω της νέας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τη δράση κατά του καρκίνου. Αυτές είναι οι απαντήσεις λοιπόν για τις ερωτήσεις 1 και 3 και τώρα θα δώσω το λόγο στη Μαρία για να απαντήσει τη δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα, η Μαρία Βιδάλα, επικεφαλής μονάδας για την ιατρική έρευνα στην ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας. Για το πρώτο σας ερώτημα, το τρίτο δηλαδή, πού είναι τα χαρτιά μου. Το εάν η Κομισιόν θα δώσει περισσότερο βάρος ε, στον ορθοκολικό καρκίνο στα μελλοντικά προγράμματα υγείας και πώς ε, θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να στηρίξουν τη διαδικασία προγραμματισμού. Όσον αφορά τις προσπάθειες ελέγχου, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία και για να έχουμε στον δυνατόν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Υπάρχουν διεθνείς προσπάθειες οι οποίες εστιάζονται σε ευρύτερα ζητήματα όσον αφορά την πρόβλεψη, παθογένεση, ε, ανείχνευση, θεραπεία και φροντίδα ασθενών. Έτσι Έχουμε φτάσει σε κατανομή 458 εκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα για τον καρκίνο που αντιπροσωπεύει γύρω στα 180 έργα με 1500 εργαστήρια που εμπλέκονται και 300 εκατομμύρια από το τωρινό πρόγραμμα πλαίσιο που μιλάμε για 75 έργα δηλαδή για την περίοδο 2007 με 2010. Όσον αφορά συγκεκριμένα τον ορθοκολικό καρκίνο. Έχουμε πάνω από 62 εκατομμύρια που έχουν πάει σε συνεργασίες έρευνας υπό το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, δηλαδή 2002-2006 και 41 εκατομμύρια ευρώ αφιερώνονται τώρα, όπως είπα, σε μια τριετή περίοδο του εβδόμου προγράμματος για την έρευνα. Πάρα πολλά από αυτά τα έργα αντιμετωπίζουν απευθεία τον ορθοκολλικό καρκίνο και σχετίζονται παραδείγματο χάρη με την ε, διάγνωση από ε, διάγνωση παραγόντων κινδύνου, τον ρόλο των βλαστοκυτάρων, ε, νέα προκλινικά μοντέλα, μοριακές υπογραφές για συγκεκριμένα φάρμακα, καθώς και τρόπους βελτίωσης άλλων ε, θεραπείων όπως χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία. Αλλά στοιχεία αντιμετωπίζουν γενικότερα ζητήματα όπως την αντίσταση στη χημειοθεραπεία, τη μετάσταση ή τον ε, σχηματισμό καρκινικών ε, κιτάρων στο αίμα. Όσον αφορά τις προτάσεις για το πρόγραμμα υγείας του 2012, σκοπεύουμε να το δημοσιεύσουμε τον Ιούλιο και υπάρχουν πολλοί τομείς ε, που σχετίζονται με τον ορθοκολικό καρκίνο, αφορούν προσωπική ιατρική, δίκτες και συστήματα και μια προσέγγιση βιολογικών συστημάτων για τις ιατρικές ανάγκες επιπλέον. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό για τον προγραμματισμό του 2013 που θα δημοσιεύσουμε το 2012, η διεθνής έρευνα για τον ορθοκολικό καρκίνο θα συμπεριληφθεί επίσης και άλλοι τομείς βεβαίως. Ε, η μετάσταση, παραδείγματος χάρη, το ζήτημα του εμβολιασμού και βεβαίως νοσοποιητικές ε, θεραπείες. Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε πως ε, η Κομισιόν αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς συμμετέχουμε στο Διεθνές Consortium για το γονιδίωμα που ξεκίνησε το 2008 με ένα συνολικό φάκελο 21 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τον συντονισμό ε, μεγάλων μελετών χαρτογράφησης του γονιδιώματος του καρκίνου από διάφορους τύπους και τον καρκίνο του ορθού. Και σκοπεύουμε βέβαια να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό της έρευνας, προγραμμάτων και πολιτικών Δραστηριοποιούμαστε λοιπόν ενεργά στο συντονισμό της έρευνας μέσω ενός δικτύου αριστείας που στόχο έχει τη ε, την δικτύωση των κέντρων καρκίνου, την ε, πρωτοβουλία δηλαδή Eurocan, καθώς και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη δικτύωση εθνικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένους τομείς και υπάρχει και κάτι για τα αρχεία καρκίνου, παραδείγματος χάρη, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τυποποίηση και τις βέλτιστες πρακτικές. Και ένα άλλο για την διεθνή έρευνα, τη δικτύωση εθνικών προγραμμάτων δηλαδή, που λέγεται Transcan και ξεκίνησε επίσης φέτος. Συμμετέχουμε επίσης στην ε, πρωτοβουλία που ανέφερε ο συνάδελφος ο κ. Σρέκ, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία κατά του καρκίνου. Εμείς θα παίξουμε ε, βασικό ρόλο στον συντονισμό της έρευνας του καρκίνου και σκοπεύουμε να έχουμε συντονίσει το 1 τρίτο των ε, ερευνητικών κονδυλίων, κατά το οποίο το προσφέρει γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Όσον αφορά το μέλλον και το ερώτημά σας για το πόσο μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων του προγραμματισμού. Εμείς σκοπεύουμε στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο μόλις υιοθετήσαμε, για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και ξεκινήσαμε μια ανοιχτή διαβούλευση που είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Μαΐου και ευχαρίστως ε, να μας πούν οι ενδιαφερόμενοι Ποιο θα είναι ο καλύτερο τομέα για να επενδύσουμε στην έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο κύριος θέλω να σα ευχαριστήσω και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Η καλύτερη απάντηση είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ νομίζω. Γνωρίζω ότι είναι ώρα για βραδινό και όχι για περισσότερες ερωτήσεις, αλλά έχω να θέσω τα εξής ερωτήματα. Μιλήσατε για τη συγχρηματοδότηση ε, φορέων που συνδέονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα θέματα του καρκίνου. Στις 2 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε οργανώσει μια συζήτηση όπου αναφέρθηκε το θέμα της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού φορέα για την έρευνα για τον καρκίνο που θα συντόνιζε τις ερευνητικές δραστηριότητες αυτού του είδους. Το ερώτημά μου είναι θα ήθελε η Κομισιόν να σκεφτεί για την πρωτοβουλία αυτή και να τη βοηθήσει να ορθοποδήσει. Και κατά δεύτερον προβλέπει η Κομισιόν να πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τον ε, καρκίνο του ορθού και του παχαίου σεντέρου, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτού του καρκίνου να δώσει παραδείγματος χάρη στη δημοσιότητα ε, που να εξηγούν στον πληθυσμό την, ε, τα ωφέλη από την ανείχνευση του ορθοκολικού καρκίνου και τα μέτρα πρόληψης τα οποία θα αύξαναν τον αριθμό των ατόμων οι οποίοι προχωρούν σε ανείχνευση. Η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σρέκ πρέπει να σας πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την πολιτική υποστήριξη την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε για το έργο μας, γιατί ο στόχος μας είναι να κάνουμε και περαιτέρω πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη προγράμματα ανείχνευσης επί τη βάση του πληθυσμού. Χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν κάτι περισσότερο σε αυτά τα κράτη-μέλη. Για το θέμα του αν πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο ευρωπαϊκό φορέα ο οποίος θα συντόνιζε το περαιτέρω έργο για την έρευνα σε σχέση με τον καρκίνο και τα μέτρα δημόσιας υγείας που περιστρέφονται γύρω τον καρκίνο, νομίζω καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ εδώ να δεσμεύσω την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Είναι φανερό ότι η δημιουργία ενός νέου φορέα θα είχε και πολιτικό χαρακτήρα και θα ήταν μια φιλόδοξη ενέργεια ε, μέσα στο τωρινό πλαίσιο και μάλλον η τάση είναι ε, <clears throat> ανάστροφη για να περιοριστούν οι αποκεντρωμένοι φορείς αυτή τη στιγμή. Πάντως έχει κάποια λογική αυτή η ιδέα και εγώ έχω απόλυτη κατανόηση και υποστήριξη για αυτήν την ιδέα γιατί είμαι και εγώ επιστήμον και ξέρω ότι υπάρχει προσθέμενη αξία από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το να ε, επιφορτίζουμε ε, με τα θέματα αυτά άλλους ανεξάρτητους φορείς. Και το κέντρο της Στοκχόλμης είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω εδώ και να σας πω ότι τα τμήματα της Κομισιόν που ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη συμπάθεια για την πρότασή σας. Αλλά τώρα δεν είμαι τόσο θετικό σε σχέση με το εφικτό της πραγματοποίησης μιας τέτοιας πρότασης για τις άλλες ιδέες που αναφέρατε. πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να <clears throat> εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό οι κατευθυντές γραμμές για τον ορθοκολικό καρκίνο. Θα πρέπει καταρχήν να είμαστε υπομονετικοί. Η πλήρης εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος χρειάζονται περίπου 10 χρόνια στα κράτη-μέλη. Ένα πρόβλημα είναι η μετάφραση. Έχουμε ένα έγγραφο 400 σελίδων με χίλιες σελίδες βιβλιογραφίας δεν θα ήταν εφικτό να το μεταφράσουμε αυτό το έγγραφο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο επίτομο συνοπτικό φυλάδιο που να, να παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία. Θα το σκεφτούμε αυτό. Για τα θέματα της επικοινωνίας. οι ίδιες οι κατευθυντήριε γραμμές <clears throat> περιλαμβάνουν έμεσα μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος ανείχνευσης για τον καρκίνο αυτό, ότι όλοι οι πολίτες οι οποίοι περιλαμβάνονται στη σφαίρα εφαρμογής αυτού του προγράμματος ανείχνευσης θα πρέπει να την χάνουν προσωπικής επαφής από τις αρμόδιες αρχές. Νομίζουμε ότι θα ήταν πολύ θετικό να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση, να στέλνει κανείς ένα γράμμα σε αυτά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στο πρόγραμμα αυτό και να τους ζητάει κανείς να προχωρήσουν σε ανείχνευση. Αν τώρα πέραν αυτού χρειαζόμαστε μια συνολική προσπάθεια επικοινωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια της εταιρική σχέση για τον καρκίνο. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στα χέρια των κρατών μερών διότι τα κράτη-μέλη φυσικά είναι τα αρμόδια για τα θέματα αυτά και αυτό επομένω είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί με τη βοήθεια των κρατών μελών. Εμεί χαιρόμαστε τώρα που υπάρχει αυτή η εταιρική σχέση για τον καρκίνο και ελπίζω ότι έχω απαντήσει. Okay, thank you very much. We, uh, then... Ευχαριστούμε. Κλείνουμε αυτό το σημείο. Και περνάμε στο επόμενο που είναι μια προφορική ερώτηση για την Ασπαρτάμι. και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές χημικές ουσίες. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο στην DG Sanko για τις γλυκαντικές ουσίες και για τα η ερώτηση αφορά την ασπαρτάμι και άλλες ε, παρόμοιες γλυκα... χημικές γλυκαντικές ουσίες ε, και κατά πόσο αυτές θα απαγορευτούν ή όχι, δεδομένων των πρόσφατων ε, ερευνών. Πρόκειται για έναν τεχνητό, μια τεχνητή γλυκαντική ουσία η οποία έχει εγκριθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 33 διαφορετικές ε, κατηγορίες τροφίμων. Η ασπαρτάμι συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των θετικό όταν αυτός θεσπίστηκε το 1994 πριν από εκείνη την ημερομηνία είχε εγκριθεί σε εθνικές νομοθεσίες. Όλες οι προσθετικές ε, ουσίες στα τρόφιμα ε, πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Τρόφιμα. Παλαιότερα αυτό γινόταν από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα. Η Ασπαρτάμι αξιολογήθηκε το 1984 για πρώτη φορά και έκτοτε έχει αξιολογηθεί ακόμα πέντε φορές. Τελευταία φορά ήταν το 2009 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ασφάλεια της ουσίας αυτής επιβεβαιώθηκε και δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς για την ουσία αυτή. Στον τομέα των προσθετικών τροφίμων ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο υιοθετήθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2008. Αυτή η νέα νομοθεσία απαιτεί ότι κάθε προσθετική ουσία συμπεριλαμβανομένων των ουσιών για τις οποίες μιλάμε θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου. Δεδομένων των επανειλημμένων αξιολογήσεων στο παρελθόν, τα κράτη-μέλη ΕΦΣΑ και η Κομισιόν δεν θεώρησαν, δεν εξέτασαν μάλλον την πλήρη ε, επαναξιολόγηση της Ασπαρτάμης ε, ως πρώτη προτεραιότητα τη στιγμή που συντάχθηκε το πρόγραμμα ε, νέων αξιολογήσεων δόθηκε προτεραιότητα σε, άλλα, σε άλλες σε προστατικές ουσίες που είχαν αξιολογηθεί παλιότερα από την Ασπαρτάμι. Και έρχομαι στις δύο νέες μελέτες όταν ε, γνωρίσαμε, είδαμε αυτές τις νέες μελέτες, στις οποίες αναφέρεται αυτή η ερώτηση, ρωτήσαμε στην την ΕΦΣΑ ε, την 1η Φεβρουαρίου για νέα αξιολόγηση και επίσης κατά πόσο οι δύο αυτές μελέτες θα απαιτούσαν την αναθεώρηση των ισχυουσών επιστημονικών απόψεων για την Ασπαρτάμι. Η ΕΦΣΑ εξέδωσε δήλωση στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δύο μελέτες δεν ε, αιτιολογούν ε, την αναθεώρηση των προηγούμενων αξιολογήσεων. Εγώ θα ήθελα να τονίσω πως η ΕΦΣΑ δούλεψε για αυτή τη δήλωση μαζί με την Γαλλική Υπηρεσία Αξιολόγησης Κινδύνου, η οποία έφτασε στην ίδια, στο ίδιο συμπέρασμα που δημοσιεύθηκε μόλις αυτή την εβδομάδα. Το Δεκέμβριο του 2010 παρουσιάστηκε η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ για την ασφάλεια των προστατικών ουσιών. Πέρα από τα όσα είπε η ΕΦΣΑ στο Φεβρουάριο, το πάνελ της ΕΦΣΑ αναλύει με λεπτομέρειες την νέα αυτή μελέτη που έκανε ένας Ιταλός επιστήμονας, ο καθηγητής ε, Φροσούτη, Στις μελέτες, στη μελέτη αυτή καθώς και στη μελέτη ε, και Ισδανέζικης Αρμόδιας Υπηρεσίας ε, φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ασπαρτάμ και στην εθανόλη. Όμως ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένε μελέτες. Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί, εντό του 2011, προβλέπεται αυτό, θα εξολογήσει η ΕΦΣΑ το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση της ασπαρτάμης και ε, θα προβεί σε αυτήν. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. η οποία συμφωνεί με αυτά που άκουσα χθε σε ένα πάνελ όπου ήταν παρουσική η κυρία Παρβάνοβα και όπου εξέφρασαν την άποψή τους εκπρόσωποι της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ο καθηγητής Σοφρίτο που ήταν εκεί ανέφερε αυτή την άποψη όπως και ο καθηγητής Alderson. Κατανοώ πολύ καλά ότι η Κομισιόν χρειάζεται περισσότερα στοιχεία εκτίμησης για να αναθεωρήσει τη στάση της. Μόλον τούτο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα εξή δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι η ημερήσια επιτρεπόμενη δόση έχει καθοριστεί επί τη βάση μελετών του 1970, μια εποχή που δεν υπήρχαν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιομηχανίας. Χθες όταν συζητήσαμε, οι εκπρόσωποι της τροφιμικής αρχής είπαν ότι πράγματι αυτό ήταν η προηγούμενη αξιολόγηση που είχε γίνει στις ΗΠΑ και η οποία είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη εκεί στις ΗΠΑ ήταν αυτή η οποία ελήφθη ως η απόλυτη αλήθεια από, την, ε, από τον φορέα που προηγήθη της ε, αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και μετά από την ίδια την Εύσα. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά μελέτη η οποία ποτέ δεν επανεξετάστηκε γίνεται ένα παιχνίδι λέγοντας ότι η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να επανεξετάσει, η Κομισιόν λέγοντας ότι αυτό έχει επανεξεταστεί στο φως των προηγουμένων μελετών. Αλλά αυτό το οποίο με απασχολεί περισσότερο δείχνει η μία από τις δύο μελέτες ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα για τις έγκυες γυναίκες και τα έμβρια. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά έχουμε την αρχή της προφύλαξης. Και εγώ αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν χρήσιμο να, όχι να πάρουμε μέτρα ρυθμιστικά, αλλά να πληροφορήσουμε τις γυναίκες που είναι έγκυες, οι οποίες καταναλώνουν προϊόντα light σε μεγάλη ποσότητα γιατί δεν θέλουν να πάρουν βάρος, προϊόντα που περιέχουν ασπαρτάμι, είτε είναι αναψυκτικά, είτε είναι γιαούρτια κτλ. Τα οποία θεωρούν ότι αλλιώς έχουν πολύ ζάχαρη, χωρίς να συμβαίνει αυτό. Μήπως να προειδοποιήσουμε τις γυναίκες αυτές να μην ε, καταναλώνουν πολύ τέτοια προϊόντα, δεδομένου ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ε, ποσότητα κατανάλωσης δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει ο πληθυσμός. Δεν ξέρω πόσα γιαούρτια, πόσα, ε, πόσες δόσεις αναψυκτικών πρέπει να καταναλώσει κανείς για να φτάσει στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση. Καταρχήν λοιπόν δεν υπάρχει σε καμία συσκευασία αυτή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση. Κανείς δεν την ξέρει, κανείς δεν κάνει κάποια σύσταση προς τις έγκυες γυναίκες για να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια αυτής της επιτρεπόμενης δόσης. Δεν νομίζω λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε 2, 3, 4, 5 χρόνια πρωτού κάνουμε κάτι για την ασπαρτάμη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν όχι να απαγορεύσετε την ε, ασπαρτάμη, δεν είναι αυτό το οποίο θέλω να ζητήσω, αλλά να υπάρχει μια πληροφόρηση τουλάχιστον για τις έγκυες γυναίκες ότι θα πρέπει να καταναλώνουν με ε, σύνεση τα προϊόντα τα οποία περιέχουν ασπαρτάμι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ λογική εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Η Σας ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στην χθεσινή ακρόαση και αναφέρατε αυτό το σημείο και στην ακρόαση χθες και εγώ ήμουν παρόν στην ακρόση και είπα τότε, ότι, σας είπα ότι στο τέλος Μαρτίου ήρθε η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και εμείς ως Κομισιόν φυσικά δεν θα το αφήσουμε μονάχα για την ΕΦΣΑ να ξανακοιτάξει αυτές τις μελέτες στους επόμενους 8 μήνες, αλλά θα κοιτάξουμε και εμείς μαζί με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών <clears throat> που συμβάλλουν ιδιαίτερα στα θέματα αυτά και θα εξετάσουμε και πάλι την, ε, τη σύσταση της ΕΦΣΑ, κάτι που δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Τώρα, για τις ε, δράσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να λάβουμε στο ενδιάμεσο διάστημα, αυτές που αναφέρατε, εγώ είμαι κάπως σκεπτικιστής για το θέμα αυτό, όπως είπα και χθε στην απάντησή μου. Η μελέτη που έγινε από το δανεικό ερευνητικό οίκο σε σχέση με την χρήση από γυναίκες πριν από τον τοκετό. Η μελέτη αυτή βασιζόταν σε μια υπόθεση η οποία δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης και απαιτούσε περαιτέρω έρευνα. Έχουμε ακόμα λοιπόν μια υπόθεση η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι δύσκολο να βασίσουμε την αρχή της πρόληψης σε μία υπόθεση. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα από τα θέματα είναι η ετικετοθεσία και η προειδοποίηση στα προϊόντα αυτά. Δεν μπορώ όμως να αναλάβω τη δέσμευση ότι θα κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα πολύ καλά, λέει η κυρία Λεπάζ, αλλά λυπάμαι ότι εγώ βλέπω τελείως διαφορετικά την αρχή της πρόληψης. Η αρχή της πρόληψης είναι ακριβώς όταν έχουμε υποθέσεις μονάχα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αν ξέρουμε, μιλάμε για την εφαρμογή της πρόληψης. Η αρχή της πρόληψης αφορά το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθόμαστε αν έχουμε μία βεβαιότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο είναι υποθέσεις. Μπορεί να έχει δίκιο αυτή η μελέτη, μπορεί να μην έχει δίκιο. Αλλά αν έχει δίκιο θα πρέπει εμείς να πληροφορήσουμε το ταχύτερο δυνατό τα άτομα τα οποία μπορεί να εμπλέκονται. Αυτή είναι η μόνη μου αίτηση σε εσά. Μήπως μπορώ να προσθέσω και εγώ ένα ερώτημα. Ένας τρόπος να εφαρμόσουμε την αρχή της ε, πρόληψης είναι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να θέσουν κάτι στην αγορά πρέπει να καταδείξουν ότι αυτό το οποίο έρχεται στην αγορά δεν εμπεριέχει κινδύνους και όχι αντίθετα να πρέπει εμείς να αποδείξουμε το ότι ε, είναι επικίνδυνο το προϊόν. Ίσως μπορείτε να σχολιάσετε τώρα αυτή την αντιμετώπιση εσείς. βάρος αποδείξεως είναι σαφές ότι είναι για αυτόν ο οποίος θέτει το προϊόν στην αγορά. Να σας εξηγήσω. Στην περίπτωση του REACH που αναφερόμασταν προηγουμένως υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι διάφορες ουσίες για να εγκριθούν. Αλλά εκεί υπάρχει ανεστραμμένη, ανεστραμμένο βάρος αποδείξεως. Εδώ έχουμε μια ουσία η οποία η οποία μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και εναπόκειται στην Κομισιόν και στους καταναλωτές να δείξουν ότι έχει επικίνδυνα, ε, μπορεί να έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Γιατί το βάρος αποδείξεως δεν είναι στην περίπτωση αυτή στα χέρια του παραγωγού και αυτός να πρέπει να αποδείξει ότι είναι άκακο και άβλαβες το προϊόν αυτό. Ναι, συμφωνώ ότι το βάρος αποδείξεως είναι πάντα με αυτό που θέλει να βάλει το προϊόν στην αγορά. Αλλά επαναλαμβάνομαι. Η ουσία αυτή έχει αξιολογηθεί πάρα πολλές φορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο εθνικό και κάθε φορά έχει βγει λάδι. Έχουν καταλήξει οι ερευνητές ότι οι επιστημονικές μελέτες δεν χρειάζονται μεταρρύθμιση σε σχέση με την αξιολόγηση ασφάλειας. Συγγνώμη λέει κυρία Λεπάζου, μήπως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε σχέση με το τι σημαίνει επανεξέταση. Τι θα πει επανεξέταση για σας. Για μένα το να επανεξετάσουμε σημαίνει να πάρουμε ένα προϊόν, να κάνουμε τις μελέτες, να δούμε αν η αξιολόγηση η οποία έχει γίνει ήταν σωστή ή όχι. Αυτό όμως το οποίο έχει γίνει στην πράξη είναι ότι υπήρξαν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει για την ασπατάμη. κάποιος τις κοίταξε και κάθε φορά είπανε, μα αυτό δεν ανατρέπει τις προηγούμενες απόψει μα. Αυτό σημαίνει για σα επανεξέταση. Κομισιόν. Όταν λέω επανεξέταση, αυτό περιλαμβάνει όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έγιναν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της περίοδου επανεξέτασης. Δεν πρόκειται για ένα μονάχα στοιχείο, αλλά για μια επανεξέταση κοιτάτε τη συνολική εικόνα στην περίπτωση της Ασπαρτάμης, όλες αυτές τις... Ε, την ουσία που εξετάζεται κάθε φορά, όχι μονάχα όχι μονάχα σε σχέση με την καρκινογόνο ενδεχόμενη λειτουργία ή τα προβλήματα για τις ε, εγγύους, αλλά γενικά. Και γι' αυτό σας λέω ότι η ΕΦΣΑ έκανε την τελευταία της επανεξέταση το 2009 και αυτό αναφέρεται σαφώς στην δήλωση της ΕΦΣΑ ότι αυτή η επανεξέταση κάλυψε όλα τα στοιχεία ακόμα και την βιβλιογραφία που δεν έχει ε, εξεταστεί από ομοτήμους, δεν έχει αναθεωρηθεί από ομοτήμους. Δεν είναι μονάχα λοιπόν η επανεξέταση μιας μελέτης, αφορά όλες τις μελέτες. Το τελευταίο το οποίο θέλω να σας πω, συμφωνώ με, ακούω αυτά που λέτε, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο είπε η ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ είπε ότι αυτό δεν είναι από τις προτεραιότητές της. Εγώ κατάλαβα ότι δεν υπήρξε κάποια επανεξέταση, επανεξιολόγηση. Μου λέτε ότι υπήρξε, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο κατάλαβα από τη χθεσινή ακρόαση. Υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας και πραγματικότητας. Μπορεί να κλείσει η Κομισιόν λοιπόν για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο και μετά πρέπει να κλείσουμε το σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι λοιπόν. Σας ξαναλέω αυτό το οποίο ε, είπα προηγουμένως. Θα συζητήσουμε αυτή την δήλωση με τα κράτη-μέλη. Θα μας πούν οι εμπειρογνώμες των κρατών μελών ποια είναι η άποψή του για αυτά που λέει η κυρία Λεπάζ και αν πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. αλλά για μένα το βασικό είναι ότι θέλω να δω την ε, αξιολόγηση της ΕΦΣΑ από το 2011 και όταν είναι διαθέσιμη θα την ξανακοιτάξουμε και θα δούμε αν πρέπει να κάνουμε νωρίτερα την επόμενη επανεξιολόγηση για την ασπατάμι, η οποία δεν επίκειται γιατί έχουμε δώσει προτεραιότητα σε άλλες ουσίες και εάν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο θα κάνουμε πιο πριν την νέα επαναξιολόγηση. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε και αυτό το σημείο. Κλείνει και τη μερίσια διάταξή μας για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 11-12 Απριλίου. Σας ευχαριστώ όλους τα μάλα.